Τα συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Συζητήσαμε δύο από τα θέματα της ημέρησιας διάταξης με την Επιτροπή ΦΑΜ. Τώρα συνεχίζουμε ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πλέον. Ξεκινάμε εγκρίνοντας την ημέρησια διάταξη. Σας ανακοινώνω ότι ο Διορισμό εκτελεστικού διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕΣ στι 9 Δεκεμβρίου. Επίσης, η συνάντηση των συντονιστών έλαβε χώρα σήμερα και ε, υιοθέτησε ορισμένε συστάσει. Ε, για την κατανομή γνωμοδοτήσεων. Αν συμφωνείτε, αύριο θα διανύμω αυτές τις, αυτή τους την έκθεση, μάλλον αυτή την κατανομή γνωμοδοτήσεων, ε, σύμφωνα με τις ε, συστάσεις που, όπως σας είπα, προέκυψαν από την Επιτροπή των, των Συντονιστών. Επίσης, θα ήθελα να εγκρίνουμε τις, τα πρακτικά συνεδριάσεων και να περάσουμε στο σημείο 5 που αφορά τη διεθνή προστασία. Κράτος μέλο υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση που υποβάλλεται από επίκο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Ναι, κυρία Βίξτρομ. Thank you, ε, Ευχαριστώ. Ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί είμαι υπεύθυνη για την αναδιατύπωση του Δουβλίνου 2. Η, προ... θέση στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε το Μάιο 2009. Έκτοτε βεβαίως ε, έχουμε... είχαμε τις εκλογές και Κοινοβούλιο και εγώ πήρα την έκθεση από την προηγούμενη συγγήτρια, την κυρία Χένις ε, Πλασέρτ. Τώρα η διαδικασία συνεχίζεται. Το Συμβούλιο πλησιάζει σε μια κοινή θέση και αναμένουμε να ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους τριμερής διάλογος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατεπήγον να σιγουρευτούμε πως η έκθεση του Κοινοβουλίου του 2009 εξακολουθεί να βρίσκει στήριξη από το νέο Κοινοβουλίο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι συμφώνησαν οι συντονιστές και έχουμε ισχυρή και ενωμένη θέση στο Κοινοβουλίο. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης χαίρομαι για το ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε θα ήθελα μάλλον η Επιτροπή να επιβεβαιώσει πως ισχύει αυτό και να μου δώσει άρα μια ισχυρή εντολή για να πάω στις διαπραγματεύσεις με βάση την έκθεση του περασμένου Μαΐου και το σημερινό αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω λοιπόν κάποια σημεία κλειδιά της έκθεσης. Μεταξύ άλλων είναι τα εξή. Μεταξύ άλλων λέω. Η αναστολή των ε, μεταφορών, ε, καθώς εμείς θεωρούμε πως πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στο τελικό έγγραφο. Επίσης υπάρχει έννοια των μελών της οικογενείας, πρόβλεψη για τους ε, ανήλικους, ε, τυχόν επαναρθώσεις και κράτηση. Μεταξύ άλλων, όπως είπα, επίσης ελπίζω πως η Φελική Προεδρία σημείωσε αυτά τα θέματα και την ε, ενωμένη θέση του Κοινοβουλίου επί της έκθεσης αυτής και ελπίζω πραγματικά η Βελγική Προεδρία να συνεργαστεί μαζί μας όταν θα πλησιάσουμε πιο κοντά στις ε, τελικές διαπραγματεύσεις επί του κειμένου. Αυτά θα ήθελα να αναφέρω πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Yes, Mrs. I was say that. Ναι, και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, σημειώνουμε την συμφωνία την οποία αναφέρατε μόλις τώρα Μας παρουσιάσατε ε, συνοπτικά το ιστορικό της υπόθεσης αυτής σε ό,τι αφορά την αδιατύπωση του Δουβλίνου 2. Ο κ. Παπα-Νικολάου ήθελε να προσθέσει κάτι πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ε, Ενδεχομένω θα μπορούσε επίση να λάβει το χώρο ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο πρώτο όμω. Πρόεδρε, θέλω μόνο να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ και να επιβεβαιώσω τα όσα είπε, ότι πράγματι συμφωνούμε με την κατεύθυνση που η ίδια μόλις ενημέρωσε το, την Επιτροπή μας και πράγματι έχουμε πολύ σημαντική εργασία να κάνουμε στη συνέχεια. Ωραία. Υπάρχει συμφωνία λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν ήθελε το λόγο. Όχι. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας, κυρία Βίστρομ. Έχω μπερδευτεί. Πήγα, ταξίδεψα σε όλε τι πόλει τη Ευρώπη, ήταν κλειστά τα αεροδρόμια. Πέρασα από Γενέβη, είμαι εξαντλημένη. Έχασα και την κάρτα μου στη κάπου και η βοηθό μου πάει να μου τη φέρει από την άλλη αίθουσα την κάρτα. Μπορούμε να κάνουμε λίγο μπλα μπλα μέχρι να έρθει. Θα το εκτιμούσα. Α, ήρθε. Όχι. Θέλετε πραγματικά να κάνω κάτι τέτοιο, λέει ο πρόεδρος. Έχετε την κάρτα εσείς. Κυρία Λάμπερτ, για να βοηθήσω τη συνάδελφο, θα κάνω λίγο μπλα μπλα για κάνα δύο λεπτά σας και όδης πολιτικής μου ομάδας ε, θέλω να πω ότι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τη θέση της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου Δεν θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα για να βρεθεί λύση στο Δουβλίνο με τα χαράς να υποστηρίξω τη θέση αυτή στο ψηφοφορία. Θέλετε να μιλήσω κι άλλο. Ο κ. Κλοντ Μωράης ε, καταφθάνει για να βοηθήσει, ο Πρόεδρος. Και εγώ να συνεχίσω με τον μπλα μπλα. Αγαπάμε την κυρία Βίξτρομ και έχασε την προηγούμενη ψηφοφορία. Υποστηρίζουμε τη θέση της, όπως την παρουσίασε. Δεν είναι, μόνο μια φράση, δεν, δεν χρονοτρίβεις αρκετά. Θα έλεγα να πάω στη δική μου ψηφοφορία, θέλω να πίσω το χρόνο αγόρευσης. Κυρία Βίκστρομ, αντί να μιλάμε τον καιρό ή να παίξουμε μουσική, ας ψηφίσουμε και να λάβουμε υπόψη. Βλέπω, βλέπω, έγκαιρα, έγκαιρα, στο τσακ. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Προχωράμε λοιπόν. Έχουν το σημείο 6. Επέκταση του πεδίου εφαρμογή για την οδηγία που αφορά τους δικαιούχους ε, διεθνούς προστασίας είναι μια συμφωνία θα ανακοίνωνα το θέμα. Η είναι και ο Σκλωτ Μωράες, έτσι δεν είναι. Θα ψηφίσουμε το προηγούμενο σημείο. Μου είπαν ακριβώ επειδή ανακοινώσατε συμφωνία, δεν, χρειαζόταν να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπω προβλεπόταν. Κύριε Μπουσουτήλ, κοιτάξτε, ο εισηγητή ζητά ψηφοφορία επικύρωση, επιβεβαίωση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο της ημερήσια διάταξη της κυρίας Βίκστρομ. Πρόεδρος, ψηφίζουμε το σημείο 5. Η κυρία Βίκστρομ είναι η συγγήτρια. Θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος. 21 υπέρ, 21, 21 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, 0 ψήφοι κατά και η κυρία Ίντφελτ δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Θα μετρήσουμε την ψήφο της υπέρ, υπέρ, θετική ψήφος. Και η κυρία Χέτο, δεν δούλεψα το μηχάνημα. Άρα 23 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία εναντίον. Ευχαριστούμε κυρία Βίκστρομ. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν, επικυρώθηκε η ψήφος. Πάμε στο σημείο 6 Άλλη μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, επέκταση του πεδίου εφαρμογή οδηγία τη σχετική με του δικαιούχου διεθνού ε, προστασία. Αυτή η συμφωνία επετεύχθη όσον αφορά την επέκταση της ε, οδηγία για την άδεια παραμονής παραμονής κλπ. Στο προηγούμενο τριμερή διάλογο έγινε στις 9 Νοεμβρίου παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βατελέτ και της Επιτρόπου Βάλστρομ. Υπάρχει και πίνακα συσχετισμών εδώ που είναι θέμα προς επίλυση σε οριζόντιο επίπεδο. Ψηφίζουμε. Πριν από αυτό, εάν συμφωνείτε, να ψηφίσουμε το κείμενο στο σύνολό του για να επιβεβαιωθεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε το Συμβούλιο. Υπάρχει λοιπόν πρόταση να ψηφίσουμε όλο στο σύνολό του το κείμενο. Ο εισηγητής ο κύριος Μωράς προτείνει λοιπόν ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου, όπως είναι στην επιστολή του Συμβουλίου του Νευρίου του 2010, για να επικυρωθεί η συμφωνία η οποία συνήφθη με το Συμβούλιο. Θέλετε το λόγο, κύριε Μωράς. Κοιτάξτε, προτείνω ψηφοφορία σε όλο το κείμενο για να μην ψηφίσουμε τρεις σελίδες. Προτείνω λοιπόν γενική ψηφοφορία, συνολική. Θα ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος, το κείμενο που ψηφίζουμε, αυτό που συμπεριλαμβάνεται στην επιστολή του Συμβουλίου του Νοεμβρίου, 18 Νοεμβρίου 2010, που είναι στο παράρτημα. Ξεκινάμε την ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Δεν δουλεύει η κάρτα. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, συν την ψήφο της κυρίας Ίντφελτ που δούλευε η κάρτα της, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά. Οπότε εγκρίνεται όλες οι υπόλοιπε τροπολογίες κατέπεσαν, οπότε πάμε στην τελική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα. Τέλος. 26, 27 υπέρ, 0 απόχες, 0 ψήφοι εναντίον, άρα εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Μουράες. Πάμε στο σημείο 7. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική αποσχόληση η είναι ο συνάδελφος ο κύριος Μωράες. Στόχος του σημείου αυτό είναι να ακούσουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της επικουρικότητας ε, που ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα μας μιλήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σμιτ θα μας παρουσιάσει την ε, πρόταση μετά θα ακούσουμε την Βελγική Προεδρία και μετά ξανά τον εισηγητή. Έχουμε όμως εδώ εκπροσώπους τεσσάρων εθνικών κοινοβουλίων. Από το Τσεχική Γερουσία, από την Αυστριακή Bundesrat, το Εθνικό Κοινοβούλιο και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπέβαλαν σχετικές γνωμοδοτήσεις, συνέβαλαν στη συζήτηση που έθεσαν το θέμα ότι δεν συνάδει αυτή η πρόταση με την αρχή της επικουρικότητας. Τους δίνουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να μιλήσουν και να εκφράσουν τη θέση των κοινοβουλίων τους. Και μετά θα μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα απαντήσει στις ανησυχίες που θα εκφραστούν. θα μιλήσει πρώτα η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Νταϊάν Σμιτ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες ε, για την πρόταση αυτή γιατί ξέρω πως υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Ελπίζω λοιπόν να διευκρινίσω κάπως τα πράγματα. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση από κοινού με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά μόνο υπόψη είναι ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει την συνθήκη Ευρωπαϊκού με τα Εθνικά Κοινοβούλια και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Εμείς προτείναμε τον Ιούλιο, όπως ξέρετε, παρουσιάσαμε αυτή την πρόταση μαζί με άλλη μία πρόταση που παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Ε, θα πρέπει να ξέρετε πως για πρώτη φορά παρουσιάζει η Κομισιόν πρόταση για μη, για ανειδίκευτους ή χαμηλά εξειδικευμένους εργάτες. Πρόκειται λοιπόν για μέρος προσπάθειας να απτυχθεί μια συνολική μεταναστευτική πολιτική και η πρόταση αυτή ανακοινώθηκε ήδη το 2005 στο σχέδιο δράση για την νόμιμη μετανάστευση. Όταν είχαμε επιλέξει να έχουμε τομεακές προσεγγίσεις. Το 2009 το πρόγραμμα της Στοκχόλμης επίσης επιβεβαίωσε την σημασία εφαρμογής ε, του σχεδίου του 2005. Οπότε η πρόταση είναι αποτέλεσμα μακροσκελών διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν με μια πράσινη βίβλο και συνεχίστηκαν ε, καθ' την προετοιμασία της πρότασης και θεωρούμε πως ε, καταλήξαμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο λαμβάνει υπόψη διαφορετικές θέσεις ε, στο σημαντικό αυτό θέμα. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως με την οικονομική κρίση δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για μετανάστες εργαζόμενους σε κάποιους τομείς ε, βραχυπρόθεσμα και αυτό συμβαίνει πράγματι, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε πως ε, μέσω μακροπρόθεσμα μια οργανωμένη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης θα συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να ανταποκριθούμε και στις δημογραφικές προκλήσεις και σε λήψη εργατικού δυναμικού. Γιατί Λοιπόν, το θεωρούσαμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ζήτηση για εποχιακούς ε, εργάτες, ε, τους χρειάζονται οι εργοδότες, ειδικά στον τομέα της γεωργίας και του τουρισμού, καθώς όλο και λιγότεροι πίκο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμοι για αυτές τις εργασίες. Ε, κατόπιν οι εποχικοί εργαζόμενοι από τρίτες χώρες χρειάζονται προστασία συχνά, γιατί συχνά αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, και εργάζονται υπό κακές συνθήκες από πλευρά υγιεινής και ασφάλειας. Ε, τέλος, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την λαθρέα μετανάστευση μέσω της νόμιμης μετανάστευσης, γι' αυτό παρουσιάσαμε αυτή την πρόταση. Οπότε η πρόταση έχει δύο βασικούς στόχους. Εισάγεται εδώ πέρα μια ειδική διαδικασία για την είσοδο και την διαμονή και η δεύτερη διαδικασία είναι να ορίσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα η πρόταση έχει 7 κυρία στοιχεία. Προβλέπει μια απλού, απλούστερες διαδικασίες και γρήγορες διαδικασίες ε, εισόδου. Έχουμε ένα όριο εισδοχής 30 ημερών, το οποίο βασίζεται σε κοινά κριτήρια όπως η ύπαρξη σύμβασης εργασίας ή προσφοράς για εργασίες με μισθό ο οποίος θα είναι τουλάχιστον ο κατώτατος. Επίσης ε, θα φορά εποχική εργασία, δηλαδή 6 μήνες το έτος. Προβλέπει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η εποχική άδεια για τρία έτη με μία διαδικασία η οποία θα διευκολύνει την επανείσοδο τα επόμενα έτη. Έχει νομικούς όρους για το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, επαφή στα κράτη-μέλη να κάνουν, να τους σε μια δοκιμασία αγοράς εργασίας και βεβαίως ε, αυτό μπορούν να το κάνουν τα κράτη-μέλη και βεβαίως οι αριθμοί είναι ξεκάθαρα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και να πω εδώ πέρα βεβαίως πως υπάρχει προτιμηση, ενωσιακή προτίμηση κάτι το οποίο σημαίνει πως ε, μπορούν να επαληθεύσουν τα κράτη-μέλη εάν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας από υπηκός της Ένωσης ή υπηκός τρίτων χωρών που κατοικούν ήδη νόμιμα στην ε, Ένωση. Επίσης απαιτείται από τους ε, εργοδότες να φροντίσουν και να αποδείξουν ότι θα υπάρχει επαρκής διαμονή. Ε, υπάρχει ένας μηχανισμός παραπώνων για τους υπηκόους τρίτων χωρών και για καθορισμένες ε, τρίτους φορείς ε, για τη διαδικασία αυτή. Δεν, προβλέπε, δεν προστίθε τώρα κάτι από πλευρά κυρώσεων, γιατί υπάρχει η συγκεκριμένη οδηγία που υιοθετήθηκε το 2009, η οποία επιβάλλει κυρώσεις ε, σε όσους απασχολούν υπηκόρους τρίτων χωρών παράνομα. Οπότε υπάρχει κάποια σύνδεση εδώ πέρα με τις κυρώσεις. Τέλος, ποια είναι τα ωφέλη της ε, πρότασης κατά την άποψή μας. Απλοί οι κανόνες ε, εισδοχής ε, των εποχιακών εργαζομένων, κάτι το σημαίνει ότι θα έρχονται πιο γρήγορα όταν τους χρειάζεται η οικονομία, λιγότεροι άνθρωποι θα δουλεύουν παράνομα σε εποχιακές εργασίες και δεν θα μένουν παραπάνω από όσο δικαιούνται. Τα άλλα βεβαίως αφορούν τις συνθήκες εργασίας για να μην υπάρχει εκμετάλλευση και να φροντίζουμε την υγεία για την ασφάλεια των ε, εποχιακών αυτών εργαζομένων και τέλος η συγκοινωνία και η κυκλική μετανάστευση από και προς τις χώρες προέλευσης, κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει πως δεν θα έχουμε και παραπάνω παραμονή, αλλά θα επιτρέψει και την ροή εμβασμάτων ε, αλλά και μεταφορά δεξιοτήτων στις χώρες αυτές, άρα θα μειωθεί η φτώχεια και θα συνεισφέρουμε στην αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Αυτή είναι μια πρώτη παρουσίαση και βεβαίω είμαι στην διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. I anticipated we should hear... Καταρχήν θα πρέπει να ακούσουμε τώρα την, ε, την Βελική Προεδρία, την ε, εισηγήτρια του Κοινοβουλίου ε, και μετά από τα μέλη των Κοινοβουλίων. Η Σαβέλ Ράις από την Βελική Προεδρία καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω με δύο λόγια το στάδιο των ασιών για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο. Όπως ε, είπε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, η πρόταση υποβλήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Το Συμβούλιο Τζάι το εξέτασε τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, η πλειοψηφία των υπουργών καλωσόρισαν αυτή την πρόταση οδηγίας, αναφέροντας ότι είναι σημαντικό να, ε, να σημειωθεί πρόοδο στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Ορισμένα σχόλια έγιναν για κάποιες από τις διατάξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας. η τεχνική εξέταση του κειμένου ε, έλαβε χώρα παράλληλα ε, στην ομάδα μετανάστευσης του Συμβουλίου από το Σεπτέμβριο, ε, η εξέταση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι θέσει των κρατών μελών δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ενώ, έχουν υποβληθεί, ενώ παραμένουν αρκετές επιφυλάξει εξέταση. Μπορούμε ήδη βέβαια να γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν, τα οποία έχουν προκύψει από αυτές τι συζητήσει. Για παράδειγμα, η διάρκεια διαμονή ε, η οποία προβλέπεται από το κείμενο ε, ε, να ανέρχεται στους 6 μήνες μέγιστο σε μια περίοδο κάθε περίοδο 12 μηνών. Υπάρχουν επιφυλάξεις γι' αυτό. Το θέμα της υποχρέωσης χορήγησης άδειας διαμονής ε, ορισμένα κράτη-μέλη αμφισβητούν αυτή την υποχρέωση και αναρωτιόνται μήπως η διαμονή θα μπορούσε να ε, γίνει επί τη βάση μιας θεώρησης. Επίσης το θέμα της ε, διάρκειας της προθεσμίας επεξεργασίας της αίτησης προβλέπεται ως 30 ημέρες ορισμένοι θεωρούν ότι είναι πολύ λίγο. Για την υποχρέωση του εργοδότη να αποδεικνύει ότι ο εργοαγαζόμενος ε, έχει ένα αξιοπρεπές κατάλημα. Ε, εδώ υπάρχουν ερωτήσεις ό,τι αφορά το τι είναι αξιοπρεπές. Μετά σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες χορήγησης ε, της, ε, ε, ε των πολιετών θεωρήσεων ή αδειών διαμονής, ε, ορισμένοι έθεσαν το θέμα της ισότητας μεταχείρισης με τους ε, ημεδαπούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ορισμένα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να συζητώνται και κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας και κατά τη διάρκεια της επόμενης ε, Προεδρίας προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Η επόμενη συνάντηση της ομάδας έχει καθοριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου, θα είναι η τελευταία επί Βελικής Προεδρίας. Η Ουγγρική Προεδρία θα συνεχίσει την εξέταση. Εμείς δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε στο δικό μας εξάμεινο την εξέταση αυτή. Είμαστε όμως στη διάθεσή σας ε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε. Merci. Now from our rapporteur, Mr. Συγητής ο κ. Μωράης τώρα έχει το λόγο. το ενδιαφέρον που δείχνουν ε, τα εθνικά κοινοβούλια, μερικά εκ των οποίων είναι παρόντα, ε, αντικατοπτρίζει την ε, πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται για ένα πακέτο περί νόμης μετανάστευσης. Για πολύ καιρό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούμε να διαχειριστούμε και το θέμα της νόμης μετανάστευσης. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται κατανοητή περιπλοκότητα του θέματος, αλλά και η ανάγκη να ρυθμίσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Το συζητήσαμε στο πρόγραμμα της Χάγης, το συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και στη Στοκχόλμη ε, και ε, έχει σχέση και με την ονοματό του κυρίου Ιακολίνο ε, και αποτελεί πακέτο ε, τμήμα ενός πακέτου προτάσεων ε, που περιλαμβάνει ε, διάφορους τρόπους νόμιμης εισόδου. Έχουμε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να, η διαμονή τους να αριθμιστεί. Στο, στην καρδιά του ζητήματος αυτού, και το είπαμε εξ αρχής, είναι το δικό μας αίτημα τίμα του Κοινοβουλίου και ομάδων του να δοθεί τέλος στην εκμετάλλευση των επιχειακών εργαζόμενων και δεύτερον ε, θέλουμε να ακολουθήσουμε μια όριμη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την είσοδο μιας ομάδας εργαζομένων που ε, κατά κάποιο τρόπο είναι παγιωμένη ως δημογραφική ομάδα. Ε, δημογραφική ομάδα εννοώ ότι έρχεται να καλύψει κάποια κενά δημογραφικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αριθμητικά στοιχεία σε ορισμένα, ορισμένα πολλά από τα κράτη-μέλη που απάντησαν αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα μόνιμο κομμάτι της οικονομίας τους. Υπάρχουν αφισβητήσεις των αριθμών, αλλά η αριθμή είναι αρκετά υψηλή. Ε, έχουμε και πολλούς παράνομους εργαζόμενους που είναι εποχιακοί εργαζόμενοι ε, και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε τις δύο αυτές πραγματικότητες, θα πρέπει να εργαστούμε πολύ όρημα για να χορηγήσουμε συγκεκριμένα δικαιώματα. Η Κομισιόν μας ε, ανέφερε ποια είναι αυτά που θεωρεί πιο σημαντικά θέματα. Για μένα η πιο σημαντική πτυχή αυτού του πακέτου είναι πρώτον να καθοριστούν οι συνθήκες και οι όροι εισόδου έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των εποχιακών εργαζομένων, εργαζομένων να εξασφαλίσουμε ε, αξιοπρεπή και οικονομική ε, ε, στέγαση και βέβαια να δούμε το θέμα των, της, των ορών εργασίας και της πληρωμής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μαζί με την Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να καθορίσουμε, να ορίσουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης ή να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην ίση μεταχείριση. Βέβαια πάντοτε κάποιοι είναι πιο ίσοι από άλλους αλλά σίγουρα στην καρδιά του ζητήματος ε, βρίσκεται ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε και είναι ποια είναι η ίση πληρωμή και ε, τι θα μπορούσε να αποτελέσει ε, κίνδυνο για τους ε, εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ημεδαπούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε από τη μια μεριά να αποφύγουμε την, την των μεταναστών, αλλά από την άλλη μεριά να αποφύγουμε επίσης να πληρώνονται πολύ λιγότερο από ε, τους εργαζόμενους Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα δικαιώματα, για παράδειγμα στο θέμα τη κοινωνική ασφάλισης που θα δοθούν σε αυτού του εργαζόμενου, ε, να δούμε του όρου εισόδου και βέβαια να καταλήξουμε σε ένα πιο σαφή ορισμό του εποχιακού εργαζόμενου. Γιατί στην πράγμα, στον πραγματικό κόσμο έχουμε συνδικάτα και επιχειρήσει ε, που ασχολούνται με το θέμα των εποχιακών εργαζομένων ε, μεταναστών και θα πρέπει να είναι σαφές για αυτούς ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι διότι εργάζονται σε κλάδους ιδιαίτερα ευαίσθητους και σημαντικούς για την οικονομία. Λοιπόν, ε, έχω να βγάλω τα εξή συμπεράσματα. Θα πρέπει να δούμε το πακέτο ως σύνολο. Δεν, δεν, δεν, δεν μπορούσαμε να δεχτούμε μια οριζόντια προσέγγιση. Έχουμε μια τομεακή προσέγγιση, αλλά αυτό ε, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να έχουμε ένα κοινό παρανομαστή. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό παρανομαστή. Ε, οι εργασίες θα είναι δύσκολες, η συζήτηση θα είναι δύσκολη, αλλά είναι πολύ χρήσιμη οι συνάδελφοι που θεωρούν πως δεν θα έπρεπε να εξετάζουμε θέματα νόμιμης μετανάστευσης ας σκεφτούν ότι ε, το, από το 1999 στη συζήτηση του Τάμπερε ε, έχουν περάσει πολλά χρόνια για να καταλήξουμε στη Λισαβόνα, όπου για πρώτη φορά ε, φτάσαμε στο σημείο να μπορούμε να ε, ρυθμίσουμε θέματα νόμιμης μετανάστευσης. Η συζήτηση θα είναι δύσκολη, το είδαν και στα Εθνικά Κοινοβούλια αυτό που προσπάθησαν να ρυθμίσουν το, το, ίδιο θέμα, αλλά είναι πολύ χρήσιμη οι, οι εκθέσεις αυτές, όλα αυτά τα κείμενα είναι πολύ σημαντικά θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να καθορίσουμε ένα σύνολο δικαιωμάτων τα οποία θα τα υποστηρίξει ευρέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μωράες. Θα ήταν δίκαιο να ακούσουμε την άποψη των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων που έθεσαν το ζήτημα της επικουρικότητας. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τόμας Γκρούλιχ εκπρόσωπος της ε, τσεχικής ε, γερουσίας. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι, η γερουσία της Τσεχίας υιοθέτησε ένα αρκετά περίπλοκο ψήφισμα που συμπεριλαμβάνει εννέα σημεία. Θα αναφέρω μόνο έξι από αυτά, τα πιο σχετικά πιστεύει η γερουσία λοιπόν η τσεχική, ότι οι συνθήκε εισόδου και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών για τους σκοπούς εποχιακή απασχόλησης είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο. Και νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης δεν χρειάζεται συνεπώ. και δεν δίνει προστιθέμενη αξία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή και τι συνέπειε και τα αποτελέσματα. Και η τσεχική γερουσία δεύτερον πιστεύει ότι αυτή η πρόταση που έγινε δεν ταιριάζει με την αρχή τη επικουρικότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της συνθήκης της Λισαβόνας και η τσεχική γερουσία υιοθέτησε αιτιολογημένη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης της Λισαβόνας και τονίζει ότι η ανάγκη να ρυθμιστεί εποχιακή ε, απασχόληση σε διάφορα κάτι μέλη, ποικίλει από χώρα σε χώρα λόγω διαφορετικών δομών των αγορών εργασίας. Πιστεύει ότι η πρόταση δεν προβλέπει αποτελεσματικό μηχανισμό που θα αποτρέπει ή των χωρών από το να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για άδεια σε άλλο κράτος μέλος αφού έχει εκνεύσει η πρώτη άδεια και έτσι αυτοί οι υπήκοοι των χωρών μπορούν να μείνουν επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πέρα του μεγίστου εξαμήνου. Και νομίζουμε ότι είναι προβληματικό να εισάγονται όροι για να δημιουργούνται συνθήκε για κυκλική, να θεσπίζονται κανόνες για κυκλική απασχόληση όπως είναι η γεωργία και ο τουρισμός, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι η φύση αυτών των επαγγελμάτων δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη, όπου η μετανάστευση χρησιμοποιείται στον οικοδομικό τομέα, Φερρυππίν. Και να αναφέρω, αναφέρω και κάποια γενικότερα συμπεράσματα, διότι η Τσεχική Δημοκρατία υιοθέτησε για πρώτη φορά τέτοια γνωμοδότηση μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα. Τα συμπεράσματά μας αναφέρονται σε εμπόδια, πραγματικά εμπόδια, του να χρησιμοποιούν τα εθνικά κράτη-μέλη το μηχανισμό των καρτών σύμφωνα με την συνθήκη της Αβώνας. Έξι γνωμοδοτήσεις τονίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα με την επικουρικότητα και τα εθνικά κοινοβούλια να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις κάρτες οδηγεί σε έλλειψη συντονισμού μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων. Και ο μικρός αριθμός των γνωμοδοτήσεων οφείλεται στο ότι τα περισσότερα κοινοβούλια δεν μπόρεσαν να σεβαστούν την χρονική περίοδο των 8 εβδομάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία IPEX, μόνο 14 κοινοβούλια μπόρεσαν να συζητήσουν την πρόταση. Ο λόγος της ελλείψης συντονισμού είναι το πώ προβλέπονται αυτέ οι κάρτε από τι συνθήκε τη Αβώνα. Έχουν περιορισμένες εξουσίε τα εθνικά κοινοβούλια να υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει την πρόταση. Οπότε αποθαρρύνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Και δεν θέλουν τόσο πολύ να συντονιστούν με άλλα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτή η οδηγία είναι ένα καλό παράδειγμα χαμένων ευκαιριών για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά η κίτρινη κάρτα και λυπούμεθα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τώρα το Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστρίας, τον κύριο Χάνες Βένιγκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε την ε, επικριτική στάση του Αυστριακού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως ε, η Κομισιόν ε, πριν από λίγες ημέρες επένεσε την αυστριακή πολιτική στον τομέα της αγοράς εργασίας αναφέροντας πως καταφέραμε να μην έχουμε μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις από την κρίση και σε όλους τους σχετικούς δείκτες η Αυστρία βρίσκεται στην κορυφή. Βεβαίως έχει και η Αυστρία ανάγκη εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι όμως ε, ε, έρχονται με βάση τις ισχύουσες ε, διατάξεις και αυτό γίνεται πράγματι όταν δεν μπορούν να καλυφθούν από υπηκόους της Ένωσης. Έτσι, δεν έχουμε το φαινόμενο να έχουμε εκμετάλλευση ανθρώπων εκτός της Ένωσης για να μειωθεί ο μισθός σε συγκεκριμένους ε, κλάδους. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 7.500 εποχιακούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες, κυρίως στον τουρισμό, την ε, γεωργία και σε κάποιες βοηθητικές εργασίες. Κατά την άποψή μας θεωρούμε πως θα έπρεπε να ισχύσει η αρχή της κοινοτική προτίμησης, δηλαδή να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες με υπηκούς της ε, κοινότητας και μην ξεχνάμε πως ε, το 2011 ή 2014 θα εκπνεύσει η ε, σχετική ρύθμιση για την ε, μεταβατική περίοδο. Επίσης, η εκπρόσωπο... για αυτά τα οποία είπε η εκπρόσωπος Κομισιόν, θα ήθελα να φέρω τρία σύντομα επιχειρήματα για την δική μας θέση, για το γιατί θεωρούμε πως δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα θέμα, κάτι το οποίο αξιολογείται πολύ εποχιακά, τοπικά και περιφερειακά και κρίνεται αναλόγως. Επίσης όταν μιλάμε για έγκριση για παραπάνω από μία σεζόν είναι αδύνατον κάτι τέτοιο να γίνει για να ξέρουμε τι συνθήκες θα επικρατούν σε ε, επόμενα χρόνια. Δεύτερον, εάν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ένα ποσοστό μηδέν εάν δεν υπάρχει η ανάγκη εποχιακών εργαζομένων και τέλος δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη περίοδος ενός εξαμήνου αλλά να είναι ε, ανάλογη με τον χαρακτήρα της εργασίας και θεωρούμε ότι πάνω από 6 μήνες έχουμε ξεφύγει πια από την εποχιακή εργασία. Τα ζητήματα λοιπόν ε, αυτά της αγοράς εργασίας ε, είναι ζητήματα που παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και θεωρούμε από αυστηριακή σκοπιά πως δεν υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια ρύθμιση. Επίσης η εποχιακή εργασία είναι πολύ διαφορετική στα κράτη-μέλη και θα ε, υπάρχει πρόβλημα στο να λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη το καθένα το ποια είναι η εποχή στην οποία χρειάζεται και σε ποιους κλάδους χρειάζεται εποχιακούς ε, εργαζομένους. Και βεβαίως αν ε, θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περαιτέρω να τους αναλύσουμε τις απόψεις μας, είμαστε στην διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Με τώρα από την Βουλή των Λόρδων, ο Λόρδος Λόπερ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που, που κάλεσε τα Εθνικά Κοινοβούλια να λάβουν μέρος και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και το λόγο. Ε, έχοντας ακούσει τους συναδέλφους από την Τσεχική Δημοκρατία και από την Αυστρία μπορώ να σας πω ότι η δική μας άποψη είναι παρόμοια. Ε, έχουμε υιοθετήσει μια τεολογική εμένη γνώμη και λέμε το εξή ότι η ανάγκη για εποχιακούς εργαζόμενους είναι κοινή, ανάγκη, είναι κοινή σε πολλά στα περισσότερα κράτη-μέλη αλλά τα κράτη-μέλη διαφέρουν μεταξύ τους γιατί διαφέρουν, ε, χρειάζονται διαφορετικό αριθμό εργαζομένων για διαφορετική περίοδο, για διαφορετικό αντικείμενο κλπ. Επίσης υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη που ε, έχουν ανάγκη εργαζομένων από από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες άλλες βασίζονται πιο πολύ σε αλλοδαπού από τρίτες χώρες. Το άρθρο 79 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναγνωρίζει ότι ε, η, ο όγκο, ο αριθμός των μεταναστών, των αρπαχιακών εργαζόμενων που γίνονται δεκτοί ε, είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Ε, το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ρυθμίζεται και μπορεί να ρυθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη ε, την εθνική πολιτική και τις εθνικές ανάγκες. Η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη. Η Επιτροπή, όπως είπε, δίνει τέσσερις λόγους ε, για, μέσω των οποίων δικαιολογεί την, αρχή, την εφαρμογή της αρχής επικριτικότητας. Πρώτον, ότι η αποφάση των ενός κράτους μέλους μπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να διαστρεβλώσει, να στρεβλώσει τις μεταναστευτικές ροές. Ε, ένα κράτος ε, μέλος μπορεί να δίνει ε, τους, να δέχεται πολύ χαμηλότερους όρους και συνθήκες εργασίας και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσελκύσει πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Αυτό αφορά τους τα ελάχιστα δικαιώματα και αυτά αλλάζουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ε, δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα. Δεύτερος λόγος ε, της Κομισιόν ότι η, ε, η περιοχή Σέγγεν χρειάζεται κοινού κανόνες. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, γιατί οι κοινοί κανόνες ε, για τους νόμους μετανάστες θα μείωνε τους κινδύνους. τρίτος λόγος, ότι η εκμετάλλευση ε, και οι άσχημες συνθήκες εργασίας θα πρέπει να ε, ε, αποφευθούν μέσω ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού κειμένου. Υπάρχουν εθνικά μέτρα για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης όμως. Τελευταίος λόγος της Κομισιόν είναι ότι τον κείμενο αυτό χρειάζεται για να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες και να διευρυνθεί μια πιο παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τα ε, επιχειρήματα της Κομισιόν δεν είναι πιστικά κατά την άποψή μας. Να προσθέσω επίσης ότι ακόμα και αν υιοθετηθεί αυτή η οδηγία δεν θα εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεδομένου ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, δεν έχει επιλέξει συμμετοχή στο πρωτόκολλο 29 της συνθήκης. Αυτό όμως δεν είναι λόγος ε, για να μην εξετάσουμε εμείς ως ε, Κοινοβούλιο του Ηνωμένου αν το κείμενο αυτό συμβαδίζει με τις συνθήκες, συμμορφώνεται με τη συνθήκη. Ε, ασφαλώς και χρειάζονται <clears throat> κανόνες για την είσοδο ε, υπηκών τρίτων χωρών ως εργαζομένων και όταν μπουν χρειάζονται ε, όροι για την αξιοπρεπή τους ε, διαβίωση κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται αυτοί οι όροι και οι συνθήκες να καθορίζονται σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σούμε τώρα ξανά την εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, την κυρία Σμίτ, αν θέλει να σχολιάσει αυτά τα οποία είπαν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κυρία Σμίτ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησα ήδη σε μερικά ερωτήματα στην πρώτη μου παρέμβαση. Όμως μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά κάποια σημεία που εθίγησαν. Ακούσαμε τα Εθνικά Κοινοβούλια, λάβαμε τη γνωμοδοτήσεις τους και την επόμενη εβδομάδα θα εξετάσουμε τις γνωμοδοτήσεις θα προτιμούσαμε να έχουμε την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων στον αφάσει πρωτοβουλίε μα, όμω κατανοούμε ότι υπάρχουν και αποκλήσει απόψεων και διαφορετικέ τοποθετήσει. Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, έχουμε παραλάβει έξι αρνητικέ απαντήσει, αλλά και αρκετέ θετικέ. Και θα πρέπει να το υπογραμμίσω ότι κάποια εθνικά κοινοβούλια υποστήριξαν ε, τις προτάσεις μας, την πρότασή μας. Τώρα, Όσον αφορά διάφορα σημεία που εφήγησαν, θα ήθελα να επαναλάβω ότι αφήσαμε κάποιο περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα, όπως προανέφερα, υπάρχει η προτίμηση της Ένωσης Μπορεί να δει ποιοι είναι διαθέσιμοι στις εθνικές αγορές, αν είναι υπήκοοι της ενώσεως, της χώρας ε, και να προτιμούνται αυτοί. Και κάποιος ανέφερε τον όγκο, τον αριθμό των εργαζομένων. Ο αριθμός των υπηκών τρίτων χωρών που μπορούν να εισέλθουν είναι σαφώς καθορισμένος από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που το παγιώνει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη την κατάσταση των αγορών εργασίας στις διάφορες χώρες, στη χώρα τους και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το πώς θα οργανώσουν τις αγορές εργασίας. Μετά την προθεσμία του εξαμήνου, είναι δύσκολο ζήτημα αυτό, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη την πραγματική κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών και κάποια κράτη-μέλη επιτρέπουν σε εποχιακούς εργαζομένους να μείνουν πάνω από ένα εξάμηνο, άλλα κράτη-μέλη για συντομότερες χρονικές περιόδους. Οπότε αποφασίσαμε τελικά να κάνουμε μια πρόταση η οποία είναι ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις και προτείναμε να περιοριστεί στο εξάμεινο η διαμονή. Τόσο αφορά την κυκλική μετανάστευση, η δυνατότητα να υπάρχουν διάφορες άδειες, διαφορετικές άδειες για διάφορες εποχές, είναι κάτι σημαντικό για μας, όπως προανέφερα, διότι θα επιτραπεί και η ροή των εμβασμάτων και θα βοηθήσει την ανάπτυξη και των χωρών προέλευσης. Οπότε πρέπει να δούμε σε παγκόσμιο πλαίσιο τη μετανάστευση και στα πλαίσια της εργασίας με τίτες χώρες. Όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, γενικότερα η ανάγκη για τους εποχικούς εργοζομένους εξετάζεται από τα διάφορα κράτη-μέλη, Άλλε χώρε χρειάζονται περισσότερου εποχιακού εργαζόμενου από άλλε χώρε. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η απόφαση που λαμβάνεται από ένα κράτο μέλο ίσω να έχει συνέπειε και να επηρεάζει τα άλλα κράτη-μέλη. Κυρίω τώρα που έχουμε το χώρο Σέγγεν, χωρίς εσωτερικά σύνορα, που απαιτεί μεγαλύτερη πειθαρχία και να μειωθεί και ο κίνδυνος παρανόμων εισόδων και παράνομης διαμονής πέρα από το χρονικό όριο. Έχουμε και την οδηγία περί κυρώσεων. Να μην τη λησμονούμε, προβλέπει επιβολή κυρώσεων για εργοδότες υπηκόν τρίτων χωρών που παραμένουν παράνομα και έχουμε και την οδηγία επαναπατρισμού που θα βοηθήσει ε, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Όπως ανέφερε και ο εισηγητής ο κύριος Μωράες, αυτή η πρόταση πρέπει να ειδωθεί στα πλαίσια βρυτέρου πακέτου μαζί με άλλες οδηγίες που ήδη έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και άλλες προτάσεις που έχουν υποβληθεί, όπως η ενιαία άδεια διαμονής, Έχουμε την μπλε κάρτα, τους ε, εργαζομένους με προσόντα, με δεξιότητες. Αυτά είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν τον επόμενο χρόνο από διάφορα κάτι μέλη. Χρειάζεται ευρύτερη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε μία οδηγία που θα κάλυπτε τα πάντα. Προσπαθήσαμε αυτό να το πετύχουμε το 2001. Ήταν ανέφικτο δυστυχώς. Δεν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο. Η κατάσταση τώρα είναι διαφορετική και ελπίζω ότι με τη συναπόφαση ίσως να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, διότι τώρα και οι δύο συνομοθέτες έχουν τις ίδιες ε, εξουσίες, παρόμοιες εξουσίες. Αυτά και ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει σε Εθνικά Κοινοβούλια γραπτός, έτσι, τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για εκείνους που σήκωσαν το χέρι και ζήτησαν το λόγο. Πρώτα απ' όλα ο εισηγητής, αν έχει κάποια σχόλια, μετά από αυτά που ακούστηκαν. Πρόεδρε, ήθελα να μιλήσω τώρα πριν μιλήσουν άλλοι συνάδελφοι. Δεν φταίει η διοργάνωση των εργασιών μας, αλλά ε, είναι παράξενη η ατμόσφαιρα. Μίλησαν τα τρία κοινοβούλια και ένα κοινοβούλιο δεν, έχει, δεν συμμετέχει στην, πρόταση και άλλοι τρεις είναι κατά. Δεν παρακολουθούν συνάδελφοι προσεκτικά με την πρόταση ότι στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, η Γερμανική α, Βουλή, η Ιταλική Γερουσία και το Κοινοβούλιο, το Πολωνικό Κοινοβούλιο και η Γερουσία υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή η πρόταση δεν είναι άνευ οριμότητας και ευελιξίας. Δεν, θέλω, δεν ήθελα να υποβάλω έκθεση που δεν επιτρέπει τα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν τον αριθμό εκείνων που μπορούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια μη καινοτόμο πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματο τη κυκλική μετανάστευση, όπω αποκαλείται. Έχουμε πολυεποχιακέ άδειε καινοτομίε που δεν αντιμετωπίζονται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν τεράστιου αριθμού παράνομων μεταναστών που κάνουν εποχιακή εργασία και αυτός είναι ένας από τους θεμελιώδους λόγους για να ρυθμίσουμε την αγορά της νόμιμης μετανάστευση. Υπάρχει αυτή η παράνομη μετανάστευση και στα χώρες εκείνες που πήραν το λόγο και μίλησαν τώρα. Χρειάζεται λοιπόν ρύθμιση. Η πρόταση δεν ασχολείται άμεσα με την παράνομη εργασία. Αυτό καλύπτεται από πάλες οδηγίες και από τα ίδια τα κράτη-μέλη είναι σημαντικό να αποκατασταθεί η ισορροπία. Ποιο δηλαδή υποστήριζε την πρόταση και ποιο όχι. Ε, Βεβαίω οι επιχειρήσει και τα συνδικάτα έχουν δικά του θέματα. Ένα από αυτά ήταν ισότιμη αντιμετώπιση. Το ανέφερα αυτό. Θα υποβάλουμε αυτέ τι προτάσει και για την εποχική εργασία, οι μεταφορέ μεταξύ επιχειρήσεων και όπω το κάναμε και με την ενιαία άδεια. Και τέλο, θα θέλαμε οριζόντια πρόταση κι εμεί. Θα θέλαμε μία άδεια αλλά το Συμβούλιο ήταν κατά αυτής της προσεγγίσεως, διότι το Συμβούλιο χρόνο με το χρόνο εξακολουθούσε να μιλά για ρύθμιση της νόμης μετανάστευσης προς όφελος των πάντων, αλλά καμία πρόταση δεν υπευλήθη εκ μέρους του. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να εξετάσουμε τομεακά το ζήτημα. Ε, στο Κοινοβούλιο όμως θα εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι προτάσεις θα είναι αποδεκτές σε όλο το Κοινοβούλιο διότι άπτονται του σημαντικότατου ζητήματος της ε, παράμεση μετανάστευσης, που πολιτικό είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό για κάθε κράτο μέλο. Ευχαριστώ. Ο κ. παπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καταρχάς αμφιβολία ότι υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί εποχικοί εργαζόμενοι και ότι η Ευρώπη και πολλά κράτη-μέλη, ιδίως εκείνα που έχουν ε, μεγάλη ενασχόληση με τη γεωργία και τον τουρισμό ότι τους έχουν ανάγκη. Και βεβαίως ακριβώς επειδή πολλοί εργαζόμενοι στους τομείς αυτούς λειτουργούν παράνομα, καλός ή κακός, αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτήν την προσπάθεια που ξεκινάμε σήμερα στο ε, και στην Επιτροπή μας και αυτή την περίοδο και σε συνδυασμό βεβαίως με τις άλλες οδηγίες που ακολουθούν να εξηγήσουμε προς όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι προτιμότερο να επιλέγουν την νόμιμη οδό προκειμένου να έχουν ένα, ένα καλύτερο μέλλον και να έχουν καλύτερες ευκαιρίες ό,τι αφορά και την εργασία τους αλλά και την περαιτέρω διαβίωσή τους στα κράτη-μέλη που επιλέγουν. Βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς και, τα, και να διασφαλίσουμε ε, τα δικαιώματά τους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και ε, συμφωνώ και εγώ με τον εισηγητή μας στο θέμα αυτό. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να σκεφτεί πώς αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε για ανθρώπους που θα μείνουν σε ένα κράτος μέλος για έξι μήνες και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ε, αντίστοιχη προστασία με εκείνον που έχει μια άδεια διαμονή, που έχει μια άδεια εργασία, που εργάζεται για παράδειγμα σε ένα κράτο μέλο για πέντε χρόνια. Εκεί θέλει πολύ προσοχή. Όπω επίση ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχει οριστεί σαφώ ποιοι είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι, πώ ορίζουμε την αλλαγή των εποχών σε σχέση με του τομεί δραστηριοτήτων. Έχουμε εκεί πολλή δουλειά να κάνουμε. Απ' την άλλη πλευρά όμω, την ίδια στιγμή που θέλουμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να διασφαλίσουμε και εκεί ενδεχομένως εδράζονται και ενστάσεις από τα κράτη-μέλη, πώς δεν θα γίνει κατάχρηση αυτών των διατάξεων. Πώς δηλαδή με την ε, οδηγία που εισάγουμε δεν θα εισέλθουν κάποιοι ως εποχικοί εργαζόμενοι στα κράτη-μέλη και στη συνέχεια θα παραμείνουν εκεί παρανόμως και τελικά προσπαθώντας με την οδηγία αυτή να ε, τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να επιλέγουν την νόμιμη οδό, τελικά να έχουμε στο τέλος κατάχρηση ε, και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή από την πλευρά μας. Να είμαστε αυστηροί και να διασφαλίζουμε ότι αφού περάσει η περίοδος αυτή, όλοι οι άνθρωποι που εισήλθαν ως εποχικά εργαζόμενοι θα επιστρέψουν ε, στον τόπο τους. Για να γίνει αυτό βεβαίως πρέπει να ε, είμαστε πολύ κοντά σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τους εργοδότες, πώς δηλαδή οι εργοδότες θα παράσχουν σωστές πληροφορίες ε, και ε, βεβαίως σχέση σημαντική με αυτό έχει και η διαμονή των προσώπων αυτών, πώς θα διασφαλίζεται δηλαδή η διαμονή τους ε, την περίοδο που θα εργάζονται σε κάποιο κράτος μέλος. Σημαντικό επίσης είναι το ζήτημα της πληροφόρησης των ανθρώπων αυτών, πώς θα ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, να, να μπορούν να έχουν πληροφόρηση στη γλώσσα τους ή με βάση περιπτώσει ε, να υπάρχει δυνατότητα ε, κάποιας μετάφρασης, να, έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν τα δικαιώματά τους και σε ό,τι αφορά, ε, και σε ό,τι αφορά την περίοδο εξέτασης των αιτήσεων κλπ. Είναι δεδομένο ότι αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα με αυτό, σε αυτό το πλαίσιο και με την προσπάθεια που κάνουμε πρέπει να έχουμε αμεσότητα. Πρέπει δηλαδή κανείς να ξέρει ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για εποχικά εργαζόμενο οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες, πρέπει να είναι ε, σύντομες οι διαδικασίες για να μπορούν ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί ε, πολύ σύντομα να ε, εργάζονται στους τομείς αυτούς. Είναι δεδομένο ότι στην πορεία θα έχουμε πολύ ε, σημαντική προσπάθεια όλοι μαζί να κάνουμε ε, βεβαίως οι παρατηρήσει των συναδέλφων μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι σημαντικέ. Οι επιφυλάξει είναι δικαιολογημένε αν σκεφτεί, και την κατα... κανείς την κατάσταση με την παράνομη μετανάστευση ε, στην Ευρώπη και ιδίως για συγκεκριμένα κράτη-μέλη που υφίστανται τεράστιες πιέσεις. Ε, πραγματικά όμως ε, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να είναι ένα βήμα προς τα εμπρός αρκεί, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και από την Επιτροπή και από τον εισηγητή μας, να αποτελέσει ένα ε, κομμάτι μιας συνολικής προσέγγισης και πολιτικής για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Κυρία έχει Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ε, να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες αυτής της οδηγίας. Θα πρέπει να συζητήσουμε το σκεπτικό της και την ανάγκη ύπαρξής της. Και το σκεπτικό είναι ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνον αυτούς που έρχονται με την μπλε κάρτα, ή με βάση εθνικά προγράμματα για ε, μετανάστες εργαζόμενους και για κατόχους ανώτατης εκπαίδευσης. Χρειαζόμαστε προγράμματα και για τους εργάτες. Η κοινωνία μας γυράσκει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε υπόψη Απ' την άλλη μεριά έχουμε κοινωνίες ε, όπου οι ανάγκες καλύπτονται από ε, υπηκόους της, ε, της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό ισχύει για τη χώρα μου και για τον, την κάτω και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν ισχύει και για άλλες χώρες. Ε, συνεπώς υπάρχει και το θέμα της ε, εκμετάλλευσης ε, μεταναστών στην ε, Νότιο Ιταλία. Πέρσι θυμάστε με τα σπεριδοειδή τι έγινε. Είχαν βρεθεί Αφρικανοί να δουλεύουν και να διαμένουν υπό πολύ κακές συνθήκες. Ήταν παράνομοι εργαζόμενοι και παράνομοι διαμένοντες. Αυτό θα πρέπει να το σταματήσουμε. Η οδηγία για τους εποχικούς ε, εργαζόμενους είναι ένα πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται νομοθεσία έτσι ώστε να δώσουμε ευκαιρία στους ε, μη δικευμένους εργαζόμενους να διαμένουν στην, ε, στις χώρες μας νόμιμα. Θυμηθείτε τους ε, Αφρικανούς ε, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ισπανίας, στη Θέουτα, τη Μελίγια και θα ήθελαν να εργάζονται νόμιμα στην ε, Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα επικορικότητας. <clears throat> Αν δούμε τη συμφωνία της, του Τάμπερε, της Χάγης και της Στοκόλμης, πολλές ε, κυβερνήσεις ήδη έχουν προσυπογράψει τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Συνεπώς ε, <laughs> αναρωτιέμαι αν τα ίδια επιχειρήματα θα χρησιμοποιηθούν ε, και για, τους, ε, για την νόμιμη μετανάστευση ειδικευμένων εργαζομένων ή ισχύουν μόνο για τους ανειδικευτούς ή λίγο ειδικευμένους. Κατά μου λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα επίσης και για την ρύθμιση της κυκλικής μετανάστευσης. Σίγουρα δεν λύνουμε το πρόβλημα των εθνικών εργαζομένων. Ε, δεν πρόκειται για εποχικούς εργαζόμενους, αλλά είναι ένα θέμα διότι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι επίσης ευάλωτοι. Ίσως είναι το δεύτερο βήμα. Θα ήθελα η οδηγία αυτή να δώσει την ευκαιρία επίσης στου ε, συγκεκριμένους μετανάστες να κάνουν καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μπορεί κάποιο να ξεκινήσει ως εποχικός εργαζόμενος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εκεί θα τελειώνει και η ευρωπαϊκή του καριέρα. Ο κύριος Μωράη ε, θα είναι χρήσιμο να αναζητήσει ε, λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν και θα ήθελα ταυτόχρονα να πω στα εθνικά κοινοβούλια που νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα μόνοι τους ότι δεν είναι δυνατόν γιατί αυτή η μετανάστευση είναι εδώ και θα παραμείνει. Thank you very much, Chair. Please allow me to start by... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την γραμματεία που μας επέτρεψε να γίνει μια συζήτηση μια μισή ώρας για το πολύ αυτό σημαντικό θέμα γιατί κατά κανόνα πάντα βιαζόμαστε. Άρα... Δεν θέλω να δραματοποιήσω τα πράγματα, αλλά νομίζω πως η οδηγία αυτή μαζί με τις άλλες που ασχολούνται με τη μετανάστευση και το άσυλο είναι αν θέλετε ένα είδος ε, τεστ για το τι ρόλο θέλει να παίξει διεθνώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο, το οποίο ελπίζω να αντιλαμβάνεται το νόημα και για τα κράτη-μέλη, για τα Εθνικά Κοινοβούλια, για εμάς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τις κοινωνίες των πολιτών. Συνδικάτα, ΜΚΟ, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν μιλάμε μόνο για το ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για ένα πακέτο, αν και βεβαίως το κάθε νομοθεσία τη βλέπουμε χωριστά και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουμε με τη μετανάστευση. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ή είμαστε 27 κράτη-μέλη. Μπορούμε να έχουμε κοινούς κανόνες έστω και ελάχιστους για όλα τα κράτη-μέλη ή συνεχώς θα επικαλούμαστε την αρχή της επικουρικότητας για να συμπεριφερόμαστε με διαφορετικό τρόπο που προκαλεί σύγχυση εκτός των συνόρων μας. Νομίζω πως σήμερα είναι η μέρα. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα διεθνή ρόλο, αλλά γι' αυτό χρειάζεται κάποια συνοχή στη δική μας συμπεριφορά. Γι' αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία Νομίζω πως συζητήσαμε τόσο πολύ στην προηγούμενη θητεία όταν είχαμε το θέμα της επαναπρόθεσης για το ότι θα είχε μία ενιαία προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχαμε συζητήσει το θέμα των εποχιακών εργαζομένων. Είναι και θέμα δηλαδή του εάν τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Και αυτό είναι σημαντική προσθεμένη αξία. Δεν χρειάζεται να πούμε πως Εάν αυτό μείνει μόνο στα χέρια των κρατών μελών, α είμαστε ειλικρινεί, για κάποια κράτη-μέλη θα είναι προτεραιότητα, για άλλα όχι, αλλά ούτως ή άλλω η αλλω η νομοθεσία θα αλλάξει ανάλογα με τι αλλαγέ στην κυβέρνηση, είτε είναι πιο αριστερή, είτε πιο δεξιά, κεντρώα, δεν ξέρω. Νομίζω πως είναι φυσιολογικό να έχουμε κοινού κανόνε. έστω και ελάχιστου, όπω είπα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. αντιλαμβάνομαι πως στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες φωνές ε, απροθυμίας ε, εναντίον γιατί είναι και θέμα βεβαίως εθνικών κοινοβουλίων και συνδικάτων εθνικών και ευρωπαϊκών αλλά είμαστε ειλικρινείς Μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Μπορούμε να διασφαλίσουμε πως τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εποχιακών εργαζομένων θα προστατευτούν. Αλλά ταυτόχρονα να συμφωνήσουμε πως μπορούμε να ρυθμίσουμε τα των εποχιακών εργαζομένων που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό είναι απολύτω φυσιολογικό, γιατί ζούμε σε μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να παριστάνουμε πως δεν υπάρχει, όπως είπε και η Τζούντι, υπάρχει. Ο κόσμος αντιμετωπίζει απίστευτες συνθήκες γιατί δεν προστατεύεται και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και παρατηρώ πως το Συμβούλιο ανέφερε κάποια θέματα στα οποία δεν υπάρχει συμφωνία, τα οποία τα κράτη-μέλη εκφράζουν επιφυλάξει, Ελπίζω το Συμβούλιο να εργαστεί από αυτόν για να τα βελτιώσει και να βρει λύσεις. Αλλά όχι ε, για να σταματήσει την έγκριση της οδηγίας ε, ή την εφαρμογή της εάν υιοθετηθεί. Ελπίζω λοιπόν ως οι απαιτήσει αυτές πράγματι υφίστανται για την προστασία των ανθρώπων αυτών, των εποχιακών εργαζομένων δηλαδή. Θα ήθελα πράγματι το Συμβούλιο να αντιληφθεί αυτό το μήνυμα. Γιατί κατά την άποψή μου εδώ και αρκετό καιρό το Ευρωπαϊκό αυτό Κοινοβούλιο συμπεριφέρθηκε με τρόπο υπεύθυνο και έστειλε το μήνυμα πως θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ως σημαντικός διεθνής παίκτης. Και το ίδιο πρέπει να κάνει και το Συμβούλιο. Είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Γιακολίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών. Πρέπει να πω ότι αν ακολουθούσαμε αυτή την προσέγγιση θα αποδυναμωνόταν η οδηγία και δεν θα είχε νόημα. Ενώ είναι σημαντική οδηγία. Όπως υπενθύμισε ο συνάδελφος Μωράες, εγώ ήμουν εισηγητής της, άλλη της άλλης οδηγίας, της intra-corporate όπως αποκαλείται, που εντάσσεται σε την άλλη οδηγία και εκείνη σαν στόχο είχε μια είσοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες σε συσχετισμό με τις απαιτήσεις, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας των κρατών μελών. Κατά την άποψή μου δεν μπορούν να υπάρχουν συνθήκες εισδοχής εργαζομένων που να είναι τα, οι ίδιες για όλα τα κράτη-μέλη. Ένα πράγμα είναι όμως η επικουρικότητα και αρχή της επικουρικότητας και άλλο είναι να εγγυθεί καμίς μια ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά μια προβληματική μεγάλη. Από ό,τι θυμόμαστε αυτή η οδηγία ε, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2010 από το Ροζάρνο, που το γεγονότα εκεί, που ε, δεν ήταν μοναδικό γεγονός που συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και στο Άντερλεχτ, και στο Μάλμο, και στο Λονδίνο, και ε, στο Παρίσι, υπήρξαν επεισόδια και γεγονότα. Δεν υπάρχει κράτος μέλος όπου το πρόβλημα των εποχιακών εργαζομένων δεν αποτέλεσε αντικείμενο ζωή προσοχής από πλευράς μέσων ενημέρωσης. Είναι μια τομεακή προσέγγιση. Υπάρχουν υπηρεσίες του τα άτομα, δημόσιος τομέας, τουρισμός, γεωργία, όπου εκεί χρειάζεται υποστήριξη των ε, μεταναστών. Κάθε κάτω μέλος μπορεί να έχει το δικό του ε, μοντέλο κράτους προνοίας, το ιταλικό μοντέλο, το γερμανικό μοντέλο της εχικής δημοκρατίας, ο καθένας έχει το μοντέλο του. Η Αυστρία, η Αγγλία, λέει ο μιλητής, το ίδιο. Είναι ευαίσθητο το θέμα όμως και πάρα πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβάλλει το κύρος του διότι χρειάζεται διακοινοβουλευτική συνεργασία που θα είναι πηγή πλούτου προτάσεων, συνεισφοράς σημαντικής στον πολιτισμικό αυτό διάλογο και για αυτό το θέμα όπως και για το intra-corporate υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις κρατών μελών και επισημάνσεις θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να επιληθούν τα προβλήματα τόσο ώστε να υπάρξει πραγματική προστασία των εργαζομένων. Ξέρω ότι στην Ιταλία πολλοί εποχιακοί ε, εργαζόμενοι μαζεύουν τα μήλα, τα πορτοκάλια και απασχολούνται σε κυκλική ε, απασχόληση και το εξάμεινο είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, με το Συμβούλιο, τον εισηγητή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σημαντικά στην προσπάθεια για να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι εργασίες. Ευχαριστώ κύριος Μπουσετήλ, έχει το λόγο. Yes, thank you, Mr. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ΕΛΚ είναι ανοιχτό, δεκτικό εναντί νέων πρωτοβουλειών για την νόμιμη μετανάστευση. Το είπαμε αυτό και στο εκλογικό μας πρόγραμμα στις τελευταίες εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου και το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Συνεπώς θα είμαστε επικοδομητικοί. Του του οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια έθιξαν, ανέφεραν πολύ πιστικά επιχειρήματα για την αρχή της επικορικότητας. Ε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω το χαλί και να τα κρύψουμε. Ε, νομίζω αντιθέτως θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά. Η Κομισιόν ε, προσπάθησε να μας ε, ε, καθησυχάσει λέγοντας ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει εθνική ποσόστοση για τους μεταναστές τους οποίους θα δέχεται. Επίσης μας λένε ότι μπορεί να ε, επιλεγεί ε, η ε, εθνική προτίμηση. Αν λοιπόν αυτά τα δύο εξακολουθούν να ισχύουν, γιατί χρειάζεται η οδηγία. Αυτό είναι, αυτή είναι η δική μου απορία. Αν το σημαντικό που έρχεται από την οδηγία είναι ότι ε, μας αναγκάζει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις συνθήκες διαμονής και διαβίωσης, τότε αναρωτιέται κανείς γιατί δεν μπορούν αυτό οι χώρες να το πετύχουν μόνες τους χωρίς ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεπώς, η αρχή της επικουρικότητας είναι σημαντική και θα πρέπει να τύχει σεβασμού. Η Κομισιόν μας το χρωστάει να δικαιολογήσει καλύτερα τη χρήση, το Πώ η αρχή τη επικότητα γίνεται σεβαστή μέσω αυτού του κειμένου. Τα επιχειρήματά τη δεν αρκούν. Επίση, είπε ότι η οδηγία θα μπορούσε να μα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Από ό,τι καταλαβαίνω, από όσο ξέρω όμω, υπάρχουν άλλε οδηγίε που μα επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Μία από αυτέ είναι η οδηγία κυρώσεων εναντίον εργοδοτών που απασχολούν παρανόμως ε, εργαζόμενους. Αυτή η οδηγία ακόμα δεν έχει αρχίσει να ισχύει. Συνεπώς, ακόμα και, ακόμα και για αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα της εκμετάλλευσης, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ, να μην βιαστούμε να δεχτούμε ότι μέσω αυτής της οδηγίας θα τεθεί τέλος στην εκμετάλλευση. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Συνεπώς, δεν αντιτιθέμεθα, σε αυτή την οδηγία είμαστε ανοιχτοί, Απλώς δεν έχουμε πιστεί. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή, αλλά ε, θα πρέπει να πιστούμε. Και πιστεύω ότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει πείσει επαρκώς ότι την χάνει σεβασμού η αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Thank you, uh, also like point that was made by... Ο κ. Μούλτερ, να πω και εγώ ότι συμφωνώ με κάτι που ο κ. Μπουσουτήλ. Ε, πρώτη φορά ακούμε τις νόμες των Εθνικών Κοινοβουλίων. 12 κοινοβουλία από ό,τι ε, κατάλαβα διαφωνούν. Δεν είναι αρκετά για να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι αρκετά. Θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη και των υπολείπων κοινοβουλίων, γραπτός. Με αυτό τον, ε, και επίσης θα θέλαμε να δούμε και την απάντηση της ε, Κομισιόν σε όλα αυτά τα σχόλια, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να σταθμίσουμε τα πράγματα και να καταλάβουμε καλύτερα. Όλοι νομίζω πως συμφωνούμε ότι όσοι εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς, να τη χάνουν αξιοπρεπούς μεταχύνσεις ε, και να αποφεύγουμε την εκμετάλλευσή τους. Η αδυναμία της ε, πρότασης όμως είναι ότι δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε στατιστική που να δείχνει το μέγεθος του προβλήματος στα διάφορα κράτη-μέλη, πόσους, ε, πόσοι ε, εποχικοί εργαζόμενοι εργάζονται εκεί κλπ. Ε, η εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα είναι ευθύνη των κρατών μελών. Συνεπώς, αν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους παρανόμους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, ε, δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρουν με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, Συνεπώ δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα τη Κομισιόν που λέει ότι θα μα βοηθήσει αυτή η οδηγία να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη μετανάστευση. Ε, λοιπόν, λείπουν τα στατιστικά στοιχεία, λείπουν οι προβλέψει για το μέλλον, οι προβολέ μελλοντικέ. Ε, και σε ό,τι διαφορά το άλλο θέμα που το έθιξε και το Συμβούλιο, ε, ένα από του όρου είναι η αξιοπρεπή στέγαση. Ε, Ποιο είναι ο ορισμός της αξιοπρεπούς στέγασης. Ε, φαντάζομαι ότι ε, αυτή η έννοια διαφέρει από τη Φινλανδία στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ε, πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Μετά, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια <clears throat> διαμονής. Ποιο ήταν το επιχείρημα της Κομισιόν για να καθορίσει τη μέγιστη περίοδο στους 6 μήνες. Ε, είπε η Κομισιόν, άλλα κράτη-μέλη έχουν μέγιστο 8 μήνες, άλλα κράτη-μέλη 4, 4 μήνες, οπότε κατάληξαν στους 6. Επίσης, ε, ορισμένα επαγγέλματα, ορισμένοι τομεί ε, δεν χρειάζονται διαφορετικό μέγιστο. Ίσως η γεωργία έχει διαφορετικό, διαφορετικές ανάγκες από κάποιο άλλο τομέα. Συνεπώ δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα τη Κομισιόν για του 6 μήνε και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η περίοδο θα πρέπει να είναι η ίδια για όλα τα επαγγέλματα και όλου του τομεί. Αυτές είναι οι πρώτε ε, μου παρατηρήσει. Έχω πάρει και εγώ σχόλια και θετικά και αρνητικά. Ε, θα παρακολουθήσουμε με πολύ θετικό πνεύμα όλες τις ε, ε, προτάσεις, ε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να απαντηθούν και, οι κρίσεις. Ωραία. Κύριε Ρομέρο. Κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη και τη στάση τους έναντι αυτής της πρωτοβουλίας. Όπως είπε ο κ. Μπουσουτήλ, Είναι προφανές ότι τα κράτη-μέλη μπορούν από μόνο τους να ρυθμίσουν το θέμα των όρων εργασίας και να αποφύγουν ε, τα αρνητικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται. Επίσης είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμα για να γνωρίζουμε το μέγεθο και τις διαστάσει κατάσταση. Όμω, υπάρχουν και θέματα επικουρικότητα, υπά, ε, μάλλον, ε, παρόλο ότι υπάρχουν θέματα που άπτονται τη ε, επικουρικότητας, μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια καινούργια φάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, παρόλο ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, η κινητικότητα ε, που όλο και αυξάνεται μας οδηγεί όλο και πιο πολύ σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Συνεπώς θα πρέπει να έχουμε τα μέσα ε, και να καθορίσουμε τους όρους για να οργανωθεί αυτή η ενιαία αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι απόλυτα απαραίτητο στο μέλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι επαφίεται στα κράτη-μέλη ασφαλώς και επαφίεται στα κράτη-μέλη ασφαλώς. Και σίγουρα σεβόμαστε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι και οι ίδιοι θέλουν να αποτέλεσουν θεματοφύλακα των συνθηκών. Ναι, αλλά θα ήταν χρήσιμο να βοηθήσουν και την οικοδόμηση της Ευρώπης προς αυτή την κατεύθυνση που είναι τόσο σημαντική για να αποφύγουμε ε, ε υπερβάσεις στο μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση, τα ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, επαρκή αποτελεσματικότητα για να αποφύγουν ε, τις, ε, την κρίζα αγορά, θα πρέπει να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα μας, θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε στο μέλλον η κατάσταση να προσελκύσει ακόμα περισσότερη παράνομη μετανάστευση. Το θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Και αυτή είναι η προσθέμενη αξία της οδηγίας. Ότι δηλαδή μας βοηθάει να αποφύγουμε ε, την ε, ε, προσέλκυση νέων παράνομων μεταναστών μέσω της εφαρμογής συστημάτων αναξιοπρεπών. Αυτή είναι λοιπόν η προσθέμενη αξία πάνω στην οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανησυχώ λίγο από τις τοποθετήσεις κάποιων ε, συναδέλφων που θέλουν την εποχική αυτή μετανάστευση να την ε, μεταβάλουν ε, σε μία μόνιμη νόμιμη μετανάστευση και ε, ανησυχώ ιδιαίτερα για την κυρία που λέει πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις χώρες προέλευσης. Δεν είναι θέμα αναπτυξιακής βοήθειας, ούτε ασύλου, ούτε νομοποίησης κάποιου παράνομου πράγματος. Μιλάμε ξεκάθαρα για τους εποχιακούς εργαζόμενους τους οποίους θέλουμε να προσφέρουμε μια απασχόληση, στο μέτρο που υπάρχει η ανάγκη στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, Μπορεί να καλυφθεί αυτή η ανάγκη πρώτα απ' όλα από τα ευρωπαϊκά Και, εάν όχι, ή μάλλον να το πω αλλιώς, χρηματοδοτούμε μεγάλη ανεργία στα κράτη-μέλη. Μήπως μπορούμε να πούμε πως ε, θα βρούμε εκεί του ανθρώπου αντί να εισάγουμε εποχιακού εργαζόμενους. Εάν χρειαζόμαστε εποχιακού εργαζόμενου, νομίζω καλύτερο είναι πρώτα απ' όλα να δούμε μπορώ να καλύψω αυτήν την στη χώρα μου ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά να δούμε εάν μπορούμε εκτός των κρατών μελών να βρούμε κάποιον ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Εάν όμως υπάρχει πράγματι μια ανάγκη πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα και να ξεκαθαρίσουμε βεβαίως ε, πώς μιλάμε για εποχική απασχόληση, αλλά να ξεκαθαριστεί ποιες θα είναι οι συνθήκες για την εργασία και την είσοδο, ποιες θα είναι οι συνθήκες ζωής, ε, διαμονής, ε, αμοιβή και βεβαίως και οι κοινωνικές εισφορές. Και αυτά πρέπει να τα δούμε. Προς τα πού δηλαδή θα πηγαίνουν οι εισφορές εάν θα είναι δηλαδή στη χώρα στην οποία προσφέρεται η εργασία, γιατί και εκεί πέρα να ρωτήσει κανείς ε, θα νοσηλευτεί, ή εάν θα πάνε στη χώρα προέλευσης. Και βεβαίως τότε προκύπτουν από αυτό άλλα ερωτήματα. Εάν κάποιος επανέρχεται συνεχώς και εργάζεται συνεχώς επί ένα εξάμεινο, ε, θα έχει και συνταξιοδοτικά δικαιώματα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμιστεί αυτό έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί ε, να μην μείνουν ξεκρέμαστοι. Βεβαίως το θέμα είναι και το τι είναι μια εποχή τελικά ε, που κρατάει έξι μήνες και τι κάνουμε στις περιπτώσεις στις οποίες μία έγκυος εργαζόμενη έρχεται και μετά γεννάει. Πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση και για αυτές τις ε, περιπτώσεις. Δηλαδή το παιδί μετά είναι υπήκος μιας ε, χώρας ε, μέλους και δημιουργούνται μετά άλλες απαιτήσει όσον αφορά την ε, διαμονή τέτοιων εποχικών εργαζομένων γιατί βεβαίως το παιδί μετά πιθανώς θα έχει μια υπηκότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με τα ατυχήματα αν στους 5,5 μήνες κάποιος πάθει ατύχημα και χρειαστεί να παραμείνει πολύ καιρό στο νοσοκομείο, δεν μπορούμε να το πούμε μετά έληξε η περίοδος και πρέπει να φύγεις. Αλλά βεβαίως και να αποκλείσουμε από την άλλη μεριά της καταχρήσης. Τέλος. Ήδη με αυτά τα ερωτήματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά ακριβώς μιλάμε για ζήτημα επικουρικότητας ε, που πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα κρατη και δεν μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει επικουρικότητα. Αυτό παρεμβαίνει στα συστήματα κοινωνικής αρρωγής. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα κρατη και να δούμε ε, πώς θα ρυθμίσουμε τις πτυχές αυτές για όλους τους εμπλεκομένους. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, δεν προτιθέμει να μιλήσω, αλλά τελικά με στάθηκα κατά ανάγκη να μιλήσω. Τώρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σχεδόν ακούσαμε απάντηση από τα σχόλια που ακούστηκαν. Δηλαδή, προθυμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τη δική τους νομοθεσία αυτή τη στιγμή που θα εξασφάλιζε ότι εκείνοι που εργάζονται σε εποχική εργασία, στη γεωργία, τον τουρισμό, οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευση, όπω γίνεται τώρα. Τα κάτι μελη έχουν σχετικού νόμου, δεν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι, δεν κάνουν τι αναγκαίου ελέγχου τι περισσότερε φορέ, οπότε η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον τότε θα μπορεί να κυνηγήσει τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν προστατεύουν τους εποχικούς εργαζομένους. Και αυτοί οι εποχικοί εργαζόμενοι είναι και υπήκοοι τρίτων χωρών και υπήκοοι κρατών μελών. Οπότε οι βασικές απαιτήσει που θέλει να προβλέπει αυτή η οδηγία, δηλαδή να εξασφαλίσει τουλάχιστον ελάχιστο επίπεδο αμοιβή, συμβάσεις κλπ. Και αυτά είναι εποφελή και για τους ημεδαπούς. Να μην χρησιμοποιούμε πολύ φτηνά εργατικά χέρια και να υπονομεύουμε έτσι τις συνθήκες εργασίας. Ένα τμήμα του προβλήματος με την εποχιακή απασχόληση είναι και το εξής. Πολλοί θέλουν να έχουν πολύ φθηνούς εργαζομένους. Διότι έτσι και τα προϊόντα παράγονται είναι πολύ φθηνά. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να λύσουμε όμω όλα τα προβλήματα με τη συγκεκριμένη οδηγία. Υπάρχουν θέματα που ασφαλούν την κοινωνική ασφάλιση, πράγματι. Γι' αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ήδη κάνουν τα κράτη-μέλη, διότι υποθέτω ότι ήδη έχουν θεσπίσει κάποια μέτρα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, που αφορούν τη φορολόγηση, που αφορούν τα θέματα που άπτονται τη περίθαψη υγεία, τα βασικά δηλαδή δικαιώματα ασφάλιση. Ο ILO είναι σαφέστατο όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα για την κοινωνική ασφάλιση και ποια είναι και το ίδιο και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και εντό του συντονισμού τη κοινωνική ασφάλιση που έχουμε για του δικού μα υπηκόου και για του υπηκού των χωρών που διέρχονται τα σύνορα. Ετέθησαν θέματα όσον αφορά την αξιοπρεπή στέγαση και τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια επιλογή εντό οδηγία πλαισίου όπω αυτή είτε να προσπαθήσουμε να πούμε ποιε είναι οι βασικές αξίες να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Επίση, από αυτά που είδαμε και από αυτά που ακούσαμε εμεί οι ίδιοι είναι ξεκάθαρο ότι εξωπρεπή στέγαση σημαίνει ότι έχει ε, τρεχούμενο νερό, ότι σαν εργαζόμενος μπορείς να κάνεις ένα ντους, μπορείς να πληθείς, ότι μπορείς να μαγειρέψεις, να βρεις φαγητό, να έχει ένα κρεβάτι που δεν μοιράζεσαι με άλλου εργαζομένου. Δηλαδή, όταν δουλεύει ένα κοιμάται ο άλλο κλπ. και με βάρδιε. Ή να είναι πολύ στιμωγμένοι οι άνθρωποι σε μικρό χώρο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη πιστεύω ότι έχουν την κατάλληλη νομοθεσία σχετικά με το τι αποτελεί αξιοπρεπή στέγαση για εποχικού εργαζομένου. Αν δεν έχουν τέτοια νομοθεσία, θα πρέπει να ντρέπονται τα κράτη-μέλη. Και προφανώ κάτι πρέπει να γίνει. Άρα υπάρχει η προστιθέμενη αξία εντό αυτού που συζητούμε. Αποτελεί ένα τμήμα του γενικότερου συστήματο μεταναστεύσεω που όλα τα κράτη-μέλη και κυβερνήσει των κρατών μελών κατά το παρελθόν προσυπογράψαν. Κάποιοι ίσω μετάνιωσαν που οι προκάτοχοί του τα έκαναν, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει αυτό και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μεταξύ πολλών άλλων είναι ε, το, το διτό συστήματος που ανέφερε εργασία η κυρία Λοπέ. το θέμα των δικαιωμάτων είναι σημαντικό επίση, αλλά ένα κομμάτι είναι ότι μπορούμε να σπρώξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε τα δικαιώματα και οι καλές συνθήκες θα εφαρμόζονται σαν μέτρα όταν τα κράτη-μέλη τα ίδια θέλουν να το κάνουν αυτό από μόνοι τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ernst έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να φερθώ στα επιχειρήματα των Εθνικών Κοινοβουλίων και θεωρώ πως είναι σημαντικό και εδώ πέρα θέλω να παρακαλέσω ξανά να απευθυνθώ στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου να εξετάσουμε τα επιχειρήματα εκείνα τα οποία είναι θετικά και τα θεωρούν θετικά και άλλες χώρες και στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά. Θεωρώ πως πρέπει να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. Να μιλήσω για την κοινωνική ασφάλιση, θα ακολουθήσει αυτό. Μιλάμε για το στόχο πρώτα απ' όλα που, στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε. Τι πρέπει να ρυθμίσει η οδηγία, ποιο θα είναι το αντικείμενό της. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και διαπιστώνω πως έχουν όλα τα κράτη-μέλη εποχική εργασία και θέλουν να έχουν. Εντάξει, ανάλογα. Διαφέρει η τάξη μεγέθους βεβαίω. Επίσης διαπιστώνω πως αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτό είναι γεγονός. Σε όλες τις χώρες. Δεν ανάγκη να κοιτάμε μόνο την Ιταλία, όπου είχα πάει όπως ανέφερε και ο Ιταλός συνάδελφος. Σε πολλές χώρες υπάρχει αυτό το πρόβλημα της άσχημης εκμετάλλευσης. Εκτός νόμου. Και βλέπουμε πως και η εθνική νομοθεσία δεν έχει μπορέσει να φέρει την ίση μεταχείριση, να σταματήσει την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή ακριβώς το εθνικό επίπεδο έχει αποτύχει ως ένα βαθμό. Το ότι σκεφτόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινού κανόνες, ακριβώς επειδή υπάρχει έλλειμμα στο εθνικό επίπεδο, είναι κάτι καλό. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ευρωπαϊκή ρύθμιση, γιατί πρέπει να υπάρξει μεταχείριση. Στο μισθό, στις συνθήκες εργασίας και στα της υγείας βεβαίως. Και σε όσους είναι επιφυλακτικοί και λένε γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί να μην είναι σημαντικό για σας. Διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη στα κράτη-μέλη. Ε, να έχουμε λογικές ε, συνθήκες εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα. Δεύτερον, ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος. Λέτε να, μειωθεί, να μειωθεί η παρανομία. Ε, κάντε κάτι χρησιμοποιήστε το για να μειωθεί η παρανομία. Συμφωνώ. Και θα υποστηρίξω όλα όσα είπε ο κύριος Μωραές, πως χρειάζονται οριζόντιες λύσεις ε, και να τις προωθήσουμε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τους στόχους. Και δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε τι πάει να πει εποχικός εργαζόμενος. Άκουσα τα επιχείρηματα. Πως πρέπει ε, εποχικός να είναι 4-3 ε, μήνες, 8-12 ε, μήνες. Τι είναι δηλαδή η εποχική εργασία. Εξαρτάται από το χρόνο. Εξαρτάται από εργασία την οποία δεν κάνει κανένας άλλος στο κράτος μέλος. Δηλαδή κανείς άλλος δεν τις κάνει και είναι καλοί αυτοί οι άνθρωποι. πρέπει να πούμε ότι τι εννοούμε. Δεν θέλω να το αξιολογήσω. Άλλο ερώτημα. Ή εννοούμε πως είναι μόνο ε, αυτές οι δουλειές ή δεν θα πρέπει να έχουν ε, διαρκή χαρακτήρα. Θέλουν και οι εργοδότες να έχουν ανθρώπους οποίους γνωρίζουν και να ξανάρχονται οι ίδιοι. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι θέλουμε, τι εννοούμε. Αλλιώς θα μπλέξουμε πολύ άσχημα. Τι θέλουμε εμείς λοιπόν, να δημιουργήσουμε λογικές ανθρώπινες συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως εννοείται να πληρώνουν ε, κοινωνικές εισφορές ε, και εισφορές για τη σύνταξη. Ναι βεβαίως, αλλά πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τους στόχους. Τι θέλουμε να επιτύχουμε. Και νομίζω πως αφορμή ήταν αυτά τα οποία είδαμε και στην Ιταλία και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Thank Ωραία. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμέλ Ρέτσκι που εκπροσωπεί την Αλγερία εξ ονόματος των αντιπροσωπείων του Μαγκρέπ. Κύριε Ρέτσκι, έχετε το λόγο. Merci, Monsieur euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις της Επιτροπής. Έχω διαβάσει βέβαια και το σχέδιο οδηγίας. Έμαθα πολλά σήμερα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συγκράτησα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Ευρώπη ε, ανησυχεί για τις συνθήκες εργασίας των μελλοντικών ή και σημερινών εποχιακών εργαζόμενων, συνθήκες εργασίας, προστασίας της υγείας τους, στέγασης κλπ. Αλλά ανισχύει και για το μέλλον τους μετά, το, μετά τη λήξη της περίοδου, της εποχής ή της σύμβασής τους. Δεν άκουσα όμως ε, εδώ ούτε και είδα και στο σχέδιο οδηγίας ε, οτιδήποτε για τις ε, παρεμβάσεις των τρίτων χωρών. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για την νότια όχθη της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην Αλγερία και θα μπορούσα να συνεισφέρω συζήτηση το εξή. Να, θα μπορούσαμε, θα μπορούσα διμερός να συζητήσω ε, για το πώς θα μπορούσαμε εμείς να συνεισφέρουμε ε, σε αυτή την προστασία ε, και στρόπον ώστε η μετακίνηση αυτών των ζωμένων να αποβεί προς αμοιβαίο συμφέρον. Θα μπορούσα να σας να δούμε και το θέμα των ωφελών των τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά τι επενδύσει ή τη μείωση της φτώχεια κλπ. Δεν έχω βέβαια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και αριθμού, αλλά θα μπορούσα σίγουρα να πω ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να οδηγεί προς κάτι που υπάρχει προς να, να ευνοεί ένα φαινόμενο που υπάρχει ήδη σε ορισμένε χώρε. Μια αιμορραγία δηλαδή, μια απώλεια εργατικού δυναμικού στι δικέ μα χώρε. Γιατί εμεί έχουμε έξοδο μυαλών, εγκεφάλων, ε, ανθρώπους οποίου του έχουμε εκπαιδεύσει με πολύ κόστος ο προπολογισμό ε, της ε, παιδείας στη χώρα μου είναι το μεγαλύτερο κονδύλι του εθνικού μας προπολογισμού. Και παρόλα αυτά έχουμε πολλά μυαλά που φεύγουν ε, μόνιμα από τη χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να βγούμε και δύο κερδισμένοι, και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι δύο-τρεις ιδέες δικές μου. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Και εσάς και τον, κύριο, τον πρώτο κύριο Παντσέρη, ε, με τον οποίο είμαστε συνσηγητές στην ε, Μεσογειακή Ένωση, στην Ένωση της ε, Μεσογείου, για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρέτσκι. Η συζήτηση περιέλαβε πολλούς ομιλητές. Ε, ώρα να ακούσουμε την Κομισιόν, την κυρία Σμιτ καταρχήν. Θέλετε να σχολιάσετε κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι αρκετά σύντομη. Έχω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Δώσαμε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την μελέτη συνεπιών και κάναμε μια νέα έρευνα στα κράτη-μέλη για να έχουμε και άλλα στοιχεία. Οι εκτιμήσεις που έχουμε καταδεικνύουν ότι έχουμε πάνω από 100.000 υπηκός των χωρών ε, που είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Μπορώ να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην Ισπανία το 2008 είχαμε 24.800, Σουηδία 7.250, Ιταλία, φανταστείτε ότι υπήρχαν πολλοί και εκεί. Οπότε έχουμε κάποια στοιχεία βέβαια. Θα τα δώσουμε με αυτά τα στοιχεία αν παραλάβουμε στοιχεία κατά κράτη-μέλη βέβαια. Όσον αφορά του παράνομου εργαζομένου, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, να έχουμε στοιχεία. Τα στοιχεία που διαθέτουμε πιθανότατα αποτελούν ε, υποτίμηση της πραγματικής καταστάσεως. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω για μια ακόμη φορά στο θέμα της ανάγκης να υπάρξει μια οδηγία στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δούμε τη μετανάστευση στο σύνολό της θα πρέπει να υπάρχει συνεχτική προσέγγιση επανειλημμένα παρετέθη στο Στοκόλμη, Χάγη, το Τάμπερε, θα μπορούσα να φέρθω στο σύμφωνο για την ε, μετανάστευση και το άσυλο. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια Ευρώπη κλειστή που καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση, αλλά ότι επιτρέπει επίσης τους μετανάστες που χρειαζόμαστε να έρχουν εδώ και εκείνους που έχουν προσόντα και δεξιότητες, ήδη έχουμε οδηγίες σχετικά με το θέμα, αλλά θέλουμε και εκείνους που έχουν λιγότερα προσόντα, που δεν είναι ειδικευμένοι. Θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε ο εκπρόσωπος του Μαγκρέμπ. Δηλαδή, τι μπορούν να δώσουν αυτοί ε, οι μετανάστες στη χώρα καταγωγής. Ακόμα και αν είναι λιγότερο ειδικευμένοι ε, οι εργαζόμενοι που συζητάμε εδώ. Ίσως εδώ δεν έχουμε τόσο πολύ φυγή εγκεφάλου. Αυτούς που εργάζονται στον τουρισμό και στη γεωργία, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι θα δώσουν κάποια γνώση που αποκτούν εδώ, μια πρακτική εμπειρία που αποκτούν στα κράτη-μέλη και να τη μεταφέρουν όταν επιστρέφουν στη χώρα καταγωγή του. Άρα νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κέρδο κάποια υποστήριξη από εκεί. Αυτή η οδηγία, όπω έλεγα, αφήνει περιθώρια ευελιξία στα κράτη-μέλη Απ' την άλλη πλευρά προβλέπει κανόνες αρκετά αυστηρούς όσον αφορά τις συνθήκες και τα κριτήρια εισδοχής και τα δικαιώματα. Όλα αυτά θα πρέπει να ειδωθούν με το στόχο, δηλαδή να αποφύγουμε στρεβλώσεις όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, αλλά όπως και επανειλημμένα υπόθηκε, μιλάμε για ιδιαίτερη ευάλωτη ομάδα που πολύ συχνά αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης και με αυτή την πρόταση ελπίζουμε να κάνουμε ένα βήμα προς την προστασία αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ράις, εκπρόσωπος της Βελγικής Προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα υποθέτα. Αυτό με καθησυχάζει για τη συνέχεια των εργασιών. Είναι το εξής ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ είναι οι ίδιες όπως αυτές που εκφράστηκαν στο Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι όπως για κάθε μέσο πρώτη αντίδραση είναι η σύγκριση της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την εθνική πρακτική και την εθνική νομοθεσία που ισχύει. Νομίζω όμως ότι σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μετά από επανεξέταση του κειμένου και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράστηκαν εδώ που θα διαβιβάσω στο Συμβούλιο μετά από όλα αυτά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο το οποίο κείμενο θα μπορέσει να γίνει δεκτό από όλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα σε επιστρέψουμε στον κύριο Μωράη, τον εισηγητή μα, για να συνοψίσει και να ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου ε, για τις ε, συμβολέ τους ε, σε... κάτι το οποίο βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γιατί θα είναι δύσκολο γιατί αυτό το οποίο προέκυψε από 4-5 ε, από τις ε, παρεμβάσεις αυτές ήταν το προφανές. Οπότε ας πούμε το προφανές. Πρώτα απ' όλα, από το τάμπερι πριν από 11 χρόνια μιλάμε για την νόμιμη μετανάστευση για να νομοποιήσουμε την μετανάστευση για θετικά μέσα και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Οπότε ήταν αναπόφευκτο πως ε, όταν μπαίναμε στις τομεακές προσεγγίσεις, ε, δηλαδή τις ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές κτλ, ήταν μοιραίο ότι θα φτάναμε, θα έφτανε ο κόμπος στο χτενί. Και ποιος είναι ο κόμπος να δούμε κάποιους κοινού ε, μεταναστευτικούς δρόμους. Αλλά όταν ακούσαμε τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Βός κτλ, ακούσαμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Δηλαδή, αρκούν έξι μήνε μπορούμε να τα κάνουμε σωστά και πρέπει να μπούμε στι λεπτομέρειε. Αλλά ήταν μοιραίο πώ θα υπάρχουν εδώ πέρα πολιτικέ ευαισθησίε και επαναλαμβάνω πω για κάθε κράτο μέλο που μίλησε για την επικουρικότητα η πλειοψηφία το έχει δεχτεί και θέλει την πρόταση. Και γιατί, γιατί ξέρουν πως τα κράτη-μέλη δεν προστατεύουν τους εποχικούς εργαζόμενους, το ίδιο συμβαίνει και στην ε, Ιταλία Όπω το ο κ. Γιακολίνο, κάτι το οποίο αποτελεί ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει εφαρμογή νομοθεσία, διαφέρει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ω αποτέλεσμα, όπω είπε και ο συνάδελφος από το Μαγκρέπ, δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική μεταξύ ημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των αναπτυσσόμενων χωρών. Και αναπτυσσόμενε χώρε θέλουν μία νομοποίηση αυτή τη διαδικασία γιατί έχουμε πρόβλημα παράνομη μετανάστευση. Οπότε μοιραία θα αντιμετωπίζαμε μια πρόκληση. Αλλά αν δείτε την πρόταση αυτή, υπάρχει μια αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν. Ξέρω, ναι, ε, βεβαίω ο συνάδελφο είναι έμπειρο και δεν εντυπωσιάζεται από αξιολογήσει αντικτύπου. Μπορούσε να είναι και καλύτερη. Αλλά μπορούμε να δούμε και την ιστορία. Κοιτάξτε τα 11 χρόνια που έχουν περάσει από το Τάμπερε. Πόσε φορέ ε, προσπαθήσαμε να ε, επιτύχουμε την νομοποίηση. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε μετά την Λισαβόνα. Για του εποχικού, εγώ θα έλεγα πω είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε ένα λογικό πακέτο. Έχουμε δύσκολα ζητήματα, τα ανέφερε κύρια Λάμπερτ, κοινωνική ασφάλιση, το πεδίο εφαρμογή, τι είναι, ποιο είναι εποχικός εργαζόμενος. Εάν προσπαθήσουμε να ορίσουμε αυτά τα ζητήματα, νομίζω πως θα αντιληφθούμε γιατί τα περισσότερα κράτη-μέλη το θεώρησαν καλή ιδέα, αλλά ακόμα και εντός των πολιτικών ομάδων. Και πρέπει να το πω αυτό. Και εντός των πολιτικών ομάδων μας θα υπάρχουν εντάσεις. Όλες οι ΜΚΟ, τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Βέμπερ, έχουν εντάσεις. Και αυτό είναι μοιραίο. Και μιλάει, γιατί μιλάμε για πρώτη φορά για ανειδίκευτους και ημιεδικευμένους ανθρώπους. Ε, δηλαδή όταν θα φτάναμε σε αυτούς τους εργαζόμενους θα είχαμε τις δυσκολίες. Οπότε μιλάμε για την ουσία ενός πολύ ευαίσθητου ζητήματος για τους πολίτες μας. Πρώτα χαίρομαι για τις συνεισφορές των συναδέλφων. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια όριμη συζήτηση. Η σοβαρότητα με την οποία το προσέγγισαν οι συνάδελφοι δείχνει πως όλοι αντιλαμβάνονται πως μαζί με τις άλλες δύο νομοθεσίες ε, περνάμε σε μια νέα φάση πλέον μετά τη Λισαβόνα και το αντιλαμβανόμαστε όλοι και έχουμε άρα τη βάση για μια πολύ όρημη συζήτηση. Όσο προχωράει η συζήτηση θα φοβόμαστε λιγότερο αυτές τις προτάσεις αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχουν κάποια σημεία δύσκολα. Ζητώ λοιπόν να είστε ανοιχτόμυαλοι, να δείτε την πρόταση ως έχει και οπωσδήποτε θα εμφανιστούν πολλές από τις ανησυχίες που ακούστηκαν σήμερα στην έκθεσή μου. Αλλά τώρα είμαι πιο αισιόδοξο από ότι πριν γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί πολλοί μου προειδοποίησαν ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα με τους εποχικούς Οπωσδήποτε, αλλά η σημερινή συζήτηση νομίζω μας δείχνει πως υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε. Thank you, Mr. Moraes. We thank Ευχαριστώ κύριε Μωράης, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους ομιλητές αυτής της συζήτησης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, το έχουμε προβλέψει για το μέλλον. Το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης όπως σας ανέφερα έχει αναβληθεί, συνεπώς περνάμε στο σημείο 9. Θα ήθελα να καλωσορίσω την, την πρώην συνάδελφο, την κυρία Τζανίν Χάρις Πράσελτ. Καλώς ήρθατε ξανά στην Επιτροπή Λίμπε. Παίρναμε στο σημείο 9. Θα γίνει μια κοινή συζήτηση για την ακρίβεια. των σχεδίων ψηφίσματος ε, ε, που αφορούν το Λίχτενστάιν. Τρία στον αριθμό. Κύριε Χολμάιερ, παρακαλώ λίγη ησυχία αν μπορείτε. Όποιοι έχετε να πείτε κάτι, ε, παρακαλώ εκτός της αιθούσης. Ε, Χολμαέρ και Βάντεκαμπ είναι οι τρεις εισηγητές ε, των θεμάτων που αφορούν το Λιχτενστάιν. Θα τους δώσω το λόγο να παρουσιάσουν τις συστάσεις τους και μετά θα τα συζητήσουμε. Η προθεσμία για την υποβολή ε, διαδικαστικών τροπολογιών σε αυτά τα ψηφίσματα είναι η 6η, 6η Δεκεμβρίου. 6η Δεκεμβρίου. Δεν θα γίνουν δεκτές τροπολογίες ε, για το διατακτικό. Εκεί που λέει δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί ε, στην... Ε, σύναψη του πρωτοκόλου. Λοιπόν, να ακούσουμε τον πρώτο ε, εισηγητή. Ο κύριος Μπουσούτιλ αντικαθιστά την ε, κυρία Χολμάιρ. Συνεπώς θα του δώσω το λόγο. Κύριε Μπουσούτιλ. Then, Mr. Coelho... Α, ο κύριος Κοέγιο λοιπόν πρώτος ή ο κύριος Βάντεκαμπ. Οποιοςδήποτε από τους δύο. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το κεκτημένο Σέγγεν και ενδεχομένως και στα άλλα δύο κείμενα, η κατάσταση είναι σχετικά απλή. Όλοι περιμέναμε ε, όταν μπει η Ελβετία στο Σέγγεν να λυθεί και το θέμα του Λιχτενστάιν. Αυτό δεν συνέβη εξαιτία αντιρρήσεων κάποιου, κάποιου κράτου μέλου σχετικών με, με άλλα ζητήματα. Γι' αυτό χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο. Ε, οι αντιρρήσεις προέρχονται από την Σουηδία και την Γερμανία και είχαν σχέση με την ε, φοροαποφυγή. Το Λιχτενστάν είναι μια πολύ μικρή χώρα, δεν μπήκε στο Σέγγεν με την Ελβετία. Αυτό ε, είχε ως συνέπεια να χρειαστεί να δημιουργηθούν καινούργια εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί που δεν υπήρχαν. Και ε, αναμφιβόλως ε, η ένταξη του Λιχτενστάιν στη Σέγγεν ε, μπορεί να γίνει. Ε, υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι μέλη του χώρου Σέγγεν. Τίθε λοιπόν το θέμα του να δώσουμε άδεια να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες έχουν σχέση με την αξιολόγηση του Σέγγεν. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε αν το Λίχτενστάιν σέβεται όλα τα, πλήρη όλα τα κριτήρια Σέγγεν. Νομίζω ότι αυτά αποδειχθεί ότι τα τηρεί, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ε, περιμένουμε, να δώσουμε καταρχήν τη, το πράσινο φως έτσι ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία εξέταση του κεκτημένου. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το πράσινο φως. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριος Μπουσετήλ και κύριος Φαντανκάμπ. Κύριε Μπουσετήλ, πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι η Μονίκα Χολμαϊρ. Την αντικαθιστώ όμω για τη συζήτηση. θα αναφερθώ στη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσχώρηση του Λίχτενστάιν ε, για το πρωτοκόλλο του ε, Δουβλίνου και η κυρία Χολμάιερ υποστηρίζει αυτό το αίτημα, την προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη Συμφωνία του Δουβλίνου μαζί με την Ελβετία είναι κάτι ευπρόσδεκτο κατά την άποψή τη και είναι λογικό και αναγκαίο βήμα πρόοδου. Η άποψή της λοιπόν είναι θετική, καλωσορίζει την ολοκλήρωση αυτού του φακέλου, διεκπαιδεύση του φακέλου, εκκρεμούς επιμακρών και υποστηρίζει την σύναψη, την υπογραφή του πρωτοκόλου. Είναι ένα φυσικό βήμα που ακολουθεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και το ότι τώρα το Κοινοβούλιο δυνάμει της Εθήκης της Αβώνας έχει την εξουσία να εκφράσει σύμφωνη γνώμη ε, σημαίνει ότι πρέπει να την εκφράσουμε αυτή τη σύμφωνη γνώμη. Ένα τελικό σχόλιο, προσωπικό αν επιτρέπετε, υπό το φως και της παρουσιάσεως του κυρίου Βαντεκάμπ του επομένου θέματος που ακολουθήσει, είναι λίγο ηρωνικό θα έλεγα, ότι συζητούμε την συμπερίληψη της Ελβετίας σε κάποιες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι ακολουθεί το δημοψήφισμα αυτό το Σαββατοκυριακού στην Ελβετία. εδώ ανοίγουμε το δρόμο για την Ελβετία να κινηθεί μαζί μας σε εταιρική σχέση και η ανταπόκριση από αυτή τη χώρα ποια είναι. Εντελώς διαφορετική ανταπόκριση αν δει κανείς τα αποτελέσματα κάποιων ε, δημοψηφισμάτων λαϊκών που λαμβάνουν υπόψη στη χώρα. Θα ήταν παράληψη αν δεν εκφράζαμε εμεί ε, ανησυχίε για αυτά που συμβαίνουν στην Ελβετία. Κυρίω όσον αφορά αυτέ τι λαϊκές πρωτοβουλίε που δεν ανοίγουν αυτή τη χώρα, αντιθέτω ε, την κλείνουν. Thank you, Mr. We take note. Ευχαριστούμε. Τα σημειώνουμε αυτά τα οποία είπατε και τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Φαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και ευκαιρία. Θα έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε λίγα Ολλανδικά μετά τους ε, επιφανείς ε, ομιλητές που προηγήθηκαν. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την πρόταση που κάνω. Οι χώρες αυτές έχουν ε, ενταχθεί στο Σέγγεν και στο κεκτημένο Σέγγεν, οπότε θα αποτελέσουν μέρος και θα πληρώσουν μέρος των εξόδων για τα Ταμείο Εξωτερικών Συμφώνων. 30 Ιουνίου 2009 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ε, και ολοκληρώθηκαν 19 ε, Μαρτίου 2010 από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία όπως ξέρετε 1η Δεκεμβρίου 2009 ετέθη ενισχύ, μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώσει αυτές τις συμφωνίες. Και η συμβουλή μου είναι να τις εγκρίνουμε. Εγώ ως συζητητής είμαι θετικός με την ένταξη αυτών των χωρών στο Ταμείο Εξωτερικών ε, Συνόρων και σημειώνω αυτά τα οποία είπαν και οι προλαλήσαντες, ο προλαλήσας για το δημοψήφισμα στην Ελβετία. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, εάν κάποιος ε, σε αυτή την αίθουσα έχει καμία ιδέα για το τι σημαίνει αυτό για την δουβλινότητα της Ελβετίας. Δηλαδή θα στέλνουμε ανθρώπους πίσω στην Ελβετία εάν είναι η πρώτη χώρα εισόδου. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτόματη επαναπροώθηση των αλλοδαπών, δεν ξέρω αν υπάρχει κατάταξη των αλλοδαπών, αναρωτιέμαι εάν αυτό εμποδίζει την δυνατότητα του να έχουμε δεν ξέρω, ευθυγράμμιση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόσβαση σε ένα σύστημα ασύλου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο κάποια ιδέα. Ευχαριστώ κύριο Σένσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας και όδης εισηγητής για τους σοσιαλιστές, για τη σοσιαλιστική ομάδα, πρέπει να πω ότι υποστηρίζουμε τη θέση του εισηγητή των εισηγητών μάλλον και θεωρούμε να δοθεί θετική απάντηση σε αυτές τις εκθέσεις. Ευχαριστώ. I don't see any more hands being raised. Δεν βλέπω σηκώντα άλλα χέρια. Ίσως ε, θα έπρεπε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει ο εκπρόσωπος της να πάρει το λόγο. Όχι. Όχι Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανείς από τη, Γαλλική, από τη Βελική Προεδρία μάλλον. Συγγνώμη. Η κυρία Κέλλερ εκ νέου. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο θα μπορούσαν να απαντήσουν την ερώτησή μου, αν ξέρετε κάποια στοιχεία σχετικά με το ερώτημα που έθεσα. The Commission would like Θέλει η Κομισιόν να απαντήσει τώρα μέσω ή, να περιμένουμε την απάντηση κάποια άλλη στιγμή. Προτιμάτε να αναβάλλετε την απάντηση. Θα μπορούσατε να απαντήσετε γραπτό στην ερώτηση της κυρίας Κέλλερ. Ναι, Πρόεδρε, αυτό θα κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, έτσι. Ωραία. Εισηγητές, όχι. Ωραία. Αυτά. Η ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών, επαναλαμβάνω, είναι 6 Δεκεμβρίου, προθεσμία. 6 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι αν θέλετε να υποβάλλετε τροπολογίες στα ψηφίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί.